Ε, welcome everybody. Καλώς ορίσατε. Με μεγάλη μου χαρά σας αγγέλω ότι έχουμε εδώ προσκεκλημένους τέσσερις ειδικού και εμπειρογνώμονες για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα και για μας και για όλη την Ευρώπη και για το Κοινοβούλιο αλλά έχει σχέση και με την παιδεία και τον πολιτισμό των κρατών μελών. Πρόκειται για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης σε συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Δικαιοσύνη και Ιστορικών Υποθέσεων, θα σας το πω τώρα ή στα Ιταλικά, αν δεν σας πειράζει. Αυτή η ακρόαση. No, for Συμπαθάτε με, αλλά πριν αρχίσουμε πρέπει να σας ενημερώσω, συνάδελφοι, ότι για την έγκριση των συστάσεων των συντονιστών οι οποίοι συνεδρίασαν πριν από λίγο πρόκειται τις αποφάσεις αυτές να τις στείλουμε σήμερα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εάν δεν υπάρξει με το θα θεωρηθούν ότι εγκρίνονται αυτές οι αποφάσεις. Και τώρα θα συζητήσουμε για την ισοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη. Και πρέπει να ενημερωθούν και οι προσκεκλημένοι μας, αλλά το υπενθυμίζω και σε όλους σας, ότι αυτό το ζήτημα το επιλέξαμε λόγω της σημασίας του εδώ στην Επιτροπή μας. Αλλά σχετίζεται και με έκθεση της πρωτοβουλίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Η δε ψήφιση δεν θα γίνει τώρα κοντά, όπως νομίζουμε αυτές τις μέρες, αλλά στις 19 Οκτωβρίου. Πάντως είναι ευρύτερη σημασία στο ζήτημα για περισσότερες από μία επιτροπές. Και οπότε θα πρέπει και με διάφορα μέσα να συνειδητοποιήσουμε, να γνωρίσουμε τι γίνεται για να μάθουμε ποιες είναι οι αιτίες, ποιοι είναι οι τρόποι παρέμβασης για αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Και είδαμε το ότι μετά από τα γεγονότα του Παρισιού ε, υπήρξε μια απότομη συνειδητοποίηση του προβλήματος και είχαμε και άτυπη συνεργασία των Υπουργών και ολοκληρώθηκε με εκείνη την ε, διακήρυξη, δήλωση των Παρισίων όπου επαναλήφθηκαν οι αρχές της ε, ελευθερίας, της ανοχής και ανεκτικότητας μέσα από την παιδεία γιατί είναι ζήτημα το οποίο έχει σχέση και με συγκρούσεις είναι διαπολιτιστικό έχει σχέση με ε, τον εξτρεμισμό και την χρήση ένοπλης βίας από τους εξτρεμιστές και έχουμε επίσης για τους ξένους μαχητές ε, ε, και συγκρούσεις σε πολλές χώρες. Δεν είναι ζήτημα μερικών συγκεκριμένων μόνο χωρών. Οπότε το θέμα αυτό όλο ένα και περισσότερο βρίσκεται στο πολιτικό θεματολόγιο της Ευρώπης και δεν υπάρχει πολιτική ασφαλείας, ούτε πολιτική εξωτερική, ούτε πολιτική μετανάστευσης, η οποία δεν καλύπτει ε, αυτό το πρόβλημα και από πολιτιστικής πλευράς. Και το θέμα δεν είναι η σύγκρουση των πολιτισμών, αλλά το πού μπορεί να υπάρχει ένας κοινός τόπος και πώς είναι δυνατόν να ενισχύσουμε την υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Και πρόκειται όχι μόνο για την ριζοσπαστικοποίηση, αλλά και για αυτήν, για τις νέες γενιές κυρίως που μας απασχολεί. Οπότε και έτσι θα πρέπει όλοι να είμαστε ε, πιο προσεκτικοί για να καταλάβουμε τι γίνεται. Θα πρέπει να δοθούν κάποιες πολιτικές απαντήσεις. Θα πρέπει επίσης με όλους τους εμπλεκόμενους να παρασχεθεί βοήθεια και ενώ και τους διδάσκοντες και όχι μόνο αυτούς. Οπότε πέστε μας, παρακαλούμε, πώς να αντιμετωπίσουμε αυτού την πολιτική, κοινωνική ε, και θρησκευτική πρόκληση και τις αιτίε που βοηθούν στην ριζοσπαστικοποίηση και στην βία του εξτρεμισμού έχουμε τώρα το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης και πρόκλησης. Και θα πρέπει ομένως να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων για αυτό το πρόβλημα που έχει τώρα η Ευρώπη και άρα να δούμε πώς θα έχουμε καλύτερα ε, μια λύση η οποία να μην είναι διχαστική. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι ισχύει και για το διαδίκτυο όσον αφορά το πρόβλημα της ριζοσπαστικοποίησης, όπως ε, ξέρετε. Ε, και στην ε, Ιταλία έχουμε ήδη μια συμφωνία με την Γαλλία για αυτό. Αλλά και με άλλες χώρες, ούτως ώστε όπω προκύπτει από ένα έγγραφο που ήδη έχει συνταχθεί, για να δούμε το πώ τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα πρόκειται να ισχύσουν και στο διαδίκτυο, αλλά χωρίς να υπάρχει περιστολή των θεμελιωδών ελευθεριών. Να υπάρχει υπεύθυνη συμπεριφορά, αλλά και διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η βία του εξτρεμισμού που πολλές φορές πηγάζει από εκεί. Και Τονίζουμε την προσέγγιση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών από πλευράς ε, ασφάλειας, αλλά υπάρχει θέμα παιδείας και θέμα πολιτισμού. Αλλά θα πρέπει βέβαια να μην ξεχνούμε την περιπλοκότητα ε, του προβλήματος που πρέπει να αντιμετωπίσει η κοινωνία μας τώρα. Θα δώσουμε το λόγο στους ε, ειδικού, στους εμπειρογνώμονές μας. Πρώτα πρώτα δώσουμε το λόγο στην κυρία Καν. είναι η διευθύντρια του φορέα Inspire έμπνευση στο Λονδίνο. Και οι αρμοδιότητε του Ιδρύματο είναι το πώ δεν θα υπάρχουν ανισότητε των φίλων και πώ θα καταπολεμηθεί ο εξτρεμισμό. Και ακριβώ ε, δουλεύει με γυναίκε αλλά και με μαθητέ στα σχολεία. Κατόπιν ο κύριο Κρίστεσεν που είναι ανεξάρτητο σύμβουλο ε, στον κλάδο της ιστορίας και θα μας πει πώς θα πρέπει να ε, διδάσκεται η Ευρώπη στα σχολεία. Και επίσης εργάστηκε στα πλαίσια του δικτύου Euroclio και θα μας πει πώς μπορεί να είναι δυνατόν αυτό να το αντιμετωπίσουμε που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, συζήτηση που θα κάνουμε και μετά από αυτές τις δύο πρώτες παρουσιάσεις πρόκειται να έχουμε μισή ώρα με ερωταπαντήσεις. Και κατόπιν έχουμε παρουσίαση από τον κύριο Τιμπό Ντεμομπριάλ. Είναι δικηγόρος και πρόεδρος αλλά και συνειδητής του Ιδρύματος ή του Κέντρου για την Ιστορική Ασφαλεία της Γαλλίας σε σχέση με την πρόληψη ε, της ε, διάστασης της πολιτιστικής αλλά και εδαφικής και κατόπιν έχουμε να διευθυντεί από το, το, το τμήμα ελευθεριών και έκφρασης ε, των ε, μέσων της ε, UNESCO, τον κύριο Μπέργκερ. Οπότε βλέπετε ότι η σύνθεση του πάνελ είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε εδώ πέρα όλες στις πολιτικές ομάδες Οπότε όλοι θα σας ε, προσέξουν ε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα μας πείτε. Οπότε ευθύς αμέσως θα δώσουμε στην κυρία Καν το λόγο για την πρώτη εισήγηση. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή και καλησπέρα να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να σας εκθέσω τις σκέψεις μου όσον αφορά την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Συμφωνώ με όλα όσα προτείνει η γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής σας για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Σεπτεμβρίου φέτος και στην πρώτη αυτή πρόταση ε, καλούνται τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν στην πρόθεση της ε, ελευθερίας των δικαιωμάτων, ίσων ευκαιριών και το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και είναι έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει τον σεβασμό αυτών των ελευθεριών και ε, δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να γίνονται σεβαστή η πολυμορφία, η γλωσσική, η πολυστηγία και η θρησκευτική. Αλλά α επικεντρωθούμε τώρα στο σημείο 12 αυτή τη νομοθέτηση, εκεί που η Επιτροπή σα επιλέξει αναφέρει ότι τονίζει το πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο των γυναικών ή στην πρόληψη τη ε, ριζοσπαστικοποίηση στην οικογένεια. Και θεώρησα ότι αυτή είναι μια σύντομη φράση στη γνωμοδότηση. Αλλά για να δούμε τώρα γιατί είναι σημαντικό ο ρόλο των γυναικών, αλλά όχι μόνο μέσα στην οικογένεια. Επίσης θα ήθελα να εξηγήσω γιατί η χειραφέτηση και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς θα θωρακιστούμε έναντι του εξτρεμισμού. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές δεν δίνουμε την δέουσα σημασία στον ρόλο των γυναικών. Επίσης, να σας πω δύο λόγια για τον ρόλο των σχολείων και πώς ε, τα σχολεία μπορούν να θωρακίσουν τους μαθητές κατά της ε, ριζοσπαστικοποίησης, να τους μάθουν πώς να κρίνουν πως να έχουν κριτική σκέψη, να συζητούν τα ιδεολογικά και το πως να γίνονται κοινωνοί των ε, βασικών αξιών. Πολύ σημαντική η παιδεία και τα σχολεία. Όμως πριν προχωρήσω σε αυτά που σας είπα, να σας πω δύο λόγια για το ποιο είναι το έργο του φορέα που εκπροσωπώ. Ε, φορέα φορέας των πολιτών, η κυβέρνηση της χώρας μας έχει τέσσερις πυλώνες στην αντιτρομοκρατική στρατηγική προστασία, ε, δίωξη, προετοιμασία και πρόληψη. Θέλουμε με την πρόληψη να σταματήσουμε τον κόσμο να γίνεται ε, μέλος τρομοκρατικής ομάδας, να μην υποστηρίζουν την εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Ο φορέας μας ε, σε αυτό ε, επικεντρώνεται το, στο πώς θα γίνει αυτή η πρόληψη και πώς ε, η αφήγηση των εξτρεμισμών θα καταρριφθεί. Οπότε εμείς δουλεύουμε από τη βάση προς την κορυφή του Σιπίν και όχι το ανάποδο. Και επίσης ε, δουλεύουμε και μέσα στις μουσουλμανικές κοινότητες αλλά και ε, στους νόμιμους ε, φορείς και επίσημους φορείς. Οπότε νομίζω είναι σημαντική η φωνή των μουσουλμανικών οργανώσεων, ιδίω όσον αφορά την κατάρρευση κάποιων ε, βιολογιών που θέλουν να νομιμοποιήσουν το Ισλάμ σαν αποκλειστικότητα του Ισλαμικού κράτους και της Αλκάιδα. Και οπότε αυτό το οποίο γίνεται αμαυρώνουν αλλά και προκαλούν βία κατά των μουσουλμάνων. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική σημαντικό αυτό το κομμάτι της δράσης μας. Οπότε θέλουμε επίσης ε, να έχουμε έτσι κάποια, κάποια αφήγηση ε, αντίθετη με την ιδεολογία του ε, Ισλαμικού κράτους και του ΆΕΣΙΣ και, και του Αγίου κράτους αλλά και της Αλκάιντα και οπότε οι οργανώσεις των πολιτών είναι πολύ σημαντικές γιατί δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε η αστυνομία μόνο σε αυτό γιατί έχουμε θεολογικά κείμενα και θρησκευτικά κείμενα ε, ούτως ώστε να ενισχύσουν την ε, εξτρεμισμό των Ισλαμικών. Εμεί θα κάνουμε με τα ίδια κείμενα το αντίθετο. Οπότε ε, μας λένε ότι δεν γίνονται αρκετά ούτω ώστε να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους και αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές δεν υπάρχει η ηγεσία, δεν είναι οι φορείς καλά εξοπλισμένοι και επομένως θα πρέπει να δουλέψουν πολύ περισσότερο σε αυτό το μέτωπο. Ο φορέας μας που λέγεται Inspire συγκροτήθηκε το 2008 και είμαστε μια οργάνωση για το δικαίωμα των γυναικών και καταπολέμηση του εξτρεμισμού. Από τότε δουλεύουμε στα σχολεία με τους ε, δάσκαλους, με την ε, ε, αστυνομία και τοπικές αρχές και μουσουλμανικές κοινότητες και ξεκίνησα μια στρατεία το 2011 που λεγόταν Τζιχάντ, σκεφτικό πόλεμο δηλαδή, κατά τη βία. Οπότε θέλουμε πρώτα-πρώτα η λέξη Τζιχάντ να μην είναι μόνο λέξη στο στόμα των εξτρεμιστών για ε, γιατί τζιχάντ σημαίνει αγώνας για κάποιο δίκαιο και σωστό σκοπό. Γιατί την πήραν αυτή τη λέξη ε, και την χρησιμοποιούν για να τη βία. Μιλάμε για βία κατά γυναικών, κατά ανηλίκων γυναικών και αυτή η εκστρατεία μας ε, βοηθήθηκε από φορείς σε 32 χώρες ε, μας βοήθησαν επίσης και μας προέβαλαν τη New York Times, το Guardian, ε, εφημερίδες στα Εμμυράτα και άλλες χώρες και πρωταγωνίστησαν μουσουλμάνες. Επίσης δραστηριοποιούμεθα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί προβάλλουμε το πόσο η, άκρα δεξιά και το Ισλαμικό κράτος και οι δύο χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα δικτύωσης και το ιντερνετ για να στρατολογήσουν κόσμο. Επίσης είπαμε ότι ε, εκεί που εξηγούσαμε τι δεν πρέπει να κάνει ο κόσμο, είχε 45.000 χτυπήματα σε 72 ώρε από όλε τι χώρε. Οπότε έτσι είπαμε ότι θα πρέπει να καταρρύψουμε την υποκρισία και τα ψέματα του Ισλαμικού κράτου και είχαμε κάποια ε, αντίδραση και ανταπόκριση από πολλού ε, μαθητέ και εξήγησαν τη διαφορά μεταξύ Ισλάμ και εξτρεμισμού. Και είχαμε άλλη μία εκστρατεία making a stand, δηλαδή αντίσταση να προβάλλουμε αντίσταση και αυτό το κάναμε κατά του Χαλιφάτου και κατά ε, των προσπαθειών του Αλ Μπαγκδάντε Και οι μουσουλμάνες είπαμε ότι δεν θέλουμε άλλο πια να περιμένουμε τι θα κάνουν οι άντρες, θέλουμε να κάνουμε κάτι για αυτή την απειλή προς παιδιά και οικογένειές μας. Και είπαμε ότι η απόρριψη του Ισλαμικού κράτους είναι η αντίσταση που θέλουμε να προβάλλουμε και θέλουμε να καταρρύψουμε τα θρησκευτικά και πολιτικά τους επιχειρήματα και να ακουστεί η φωνή μας ε, καθαρά. Οπότε ξεκίνησε αυτή η καμπάνια αντίστασης πέρσι και μας ε, βοήθησε η Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας Τερεζά Μέη και η εφημερίδα Σαν που είναι η εφημερίδα της πωλήσει στη χώρα μας ε, προέβαλε στην, να, βλέπετε το κρατάω στην πρώτη σελίδα και έδειχνε μία μουσουλμάνα που φόρεγε ένα φερετζέ ένα ε, βέλο τέλος πάντων και ήταν η σημαία της Αγγλίας και ήθελε να πει αυτή η εικόνα ότι κανείς μπορεί να είναι και Βρετανός και μουσουλμάνος δηλαδή ε, θέλαμε να καταλήξουμε το, επιχείρημα ότι δεν μπορεί κανείς να είναι Βρετανός και μουσουλμάνος και αυτό είναι ένα μήνυμα ευμένος και προς τους δεξιούς εξτρεμιστές ε, στο κύριο άρθρο ΔΕ η εφημερίδα εξήγησε το πόσο σημαντικό είναι να καταπολεμηθεί όχι μόνο ο εξτρεμισμός αλλά και η Ισλαμοφοβία. Όταν είχαμε τρομοκρατική επίθεση στην Τινησία μα ζήτησε η εφημερίδα Σαν να γράψουμε ένα μανιφέστο κατά του μίσου. Ε, ότι δηλαδή είμαστε όλοι Βρετανοί, μουσουλμάνοι και μη μουσουλμάνοι και όλοι θέλουμε κράτος δικαίου, θέλουμε την ανοχή και ανεκτικότητα και επίση ε, καταγγέλουμε οτιδήποτε αναρτήσει γίνεται στο διαδίκτυο από του εξτρεμιστέ. Και είπαμε ότι όλοι οι μουσουλμάνοι και εμεί είναι υπέρ των αξιών που προβλήθηκαν τότε. Είναι βέβαια δεξιά εφημερίδα ε, το ΣΑΝ. Όμω αυτό που το διέδειξε με σωστέ διατυπώσει ότι δεν θα πρέπει κανεί να κουνάει το δάχτυλο, να κατηγορεί και να αποξενώνει του μουσουλμάνου και να τους θεωρεί πέμπτοφαλαγγίτες, αλλά ότι όλοι θα πρέπει να περαμηθούμε των κοινών αξιών της χώρας μας και έτσι θα νικήσουμε τους εξτρεμιστές. Όμως ε, αυτό θα πρέπει να γίνει με συνεργασία ή σε συνεργασία με τους μουσουλμάνους. Επίσης υπήρξε και ένα μήνυμα προς τους Βρετανούς που δεν είναι μουσουλμάνοι, ότι οι μουσουλμάνοι είναι αναπόσπαστο τμήμα της χώρας και τόσες εφημερίδες θέλουν να ευαισθητοποιήσουν τους μουσουλμάνους και το Ισλάμ και συγγνώμη θέλουν να, να τους αμαυρώσουν και θέλουν να τους ε, κατηγορήσουν σαν κοινότητα προβληματική. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει αυτές οι εφημερίδες να λάβουν υπόψη το παράδειγμα της σαν γιατί θέλουμε μια κουλτούρα που να δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό, την ισότητα και την αποφυγή διάκρισης. Και μόνο έτσι και χωρίς να αποξενώνουμε κάποια κοινότητα θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τον εξτρεμισμό. Και σε πλαίσια αυτής της ε, εκστρατείας του αντισταθείτε. Ε, δουλέψαμε σε 8 πόλεις σε Αγγλία, Ουαλία και είπαμε τα εξή προς τους μουσουλμάνες ότι θα πρέπει να βρουν κάποια άλλη αφήγηση κατά των εκτιμιστών να, μάθουν να αναγνωρίζουν τα σημάδια της ζωσβαστικοποίησης τους δείξαμε ποιοι ε, φορείς μπορούν να τις βοηθήσουν και ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους και μεταξύ των φορέων και κοινοτήτων και είπαμε ότι θα πρέπει οι γυναίκες να γίνουν πρωτοκόρες. Πρωτοκόρες και ένας από τους λόγους που το είπαμε αυτό είναι γιατί μπορούν να κάνουν τη διαφορά οι γυναίκες στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Ε, δεν να σταματήσουν να μισούν τους ε, ε, αυτούς που πρεσβεύουν ότι πρέπει να υπάρχει μίσος και αυτούς που ε, διαδίδουν εξτρεμιστικές ιδέες. Και έτσι λοιπόν οι γυναίκες θα είναι φύλακες των κοινοτήτων τους και θα είναι πηγή βοήθειας. Γιατί πολλές φορές τις ε, αγνοούμε. Είναι μάνες και άρα μπορούν να επισημάνουν ποιοι είναι οι ευάλωτοι. Μπορούν να αναγνωρίσουν τα πρώιμα σημάδια ριζοσπαστικοποίησης και μπορούν να μας βοηθήσουν να ε, φτιάξουμε μια ισχυρή ε, βρετανική και μουσουλμανική ταυτότητα από τη γέννηση κάποιου και μπορούν να βοηθήσουν τόσο ώστε να αντισταθούμε στην ιδεολογία την ε, ε, εξτρεμιστική και να καταλάβουμε τι θα πει το Ισλάμ τον 21ο αιώνα. Με σωστή παιδεία μπορούμε να καταπολεμήσουμε ε, την ερμηνεία που δίνουν εξτρεμιτές στον Ισλαμισμό για το μέλλον. Και είδαμε επίσης ότι όταν χειραφετούμε τις γυναίκες, οι γυναίκες είναι ακόμα πιο αποτελεσματικές στην καταγγελία του εξτρεμισμού και είναι αυτές που πιο εύκολα αναλαμβάνουν δράση. Πολλές κρατικές υπηρεσίες στην Αγγλία δεν χρησιμοποιούν τις γυναίκες, δεν συνεργάζονται ε, με τις γυναίκες. Οπότε αυτό το αρχίσει να αλλάζει, αλλά πολλές υπηρεσίες αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι για να συνεργαστούν με τις γυναίκες θα πρέπει να έρθουν σε άμεση επαφή μαζί τους και να μην περνούν από κάποιους ε, ε, τοπικούς ηγέτες που πολλές φορές ε, δεν, δεν έχουν κάποια ευθύνη και δεν έχουν εκλεγεί από τον κόσμο. Οπότε θα πρέπει να δούμε με τι στρατηγικές θα διδάξουμε τι γυναίκε, ούτω ώστε να προλάβουν και να καταπονημήσουν την ριζοσπαστικοποίηση. Επίση, βλέπουμε ότι πολλέ φορέ απειλούνται από του εξτρεμιστέ οι γυναίκε. Και το πρώτο που κάνουν οι εξτρεμιστέ όταν βρίσκονται, ε, όταν παίρνουν τα ενία, είναι να περιορίσουν τα δικαιώματα των γυναικών. Το ξέρουν αυτό οι γυναίκε. Και γι' αυτό ακριβώ η καταπολέμηση τη ριζοσπαστικοποίηση σημαίνει προστασία των, των δικαιωμάτων του. Οι Κριστόφ και Γούνταν είπαν ότι όταν ε, ε, απελευθερώνουμε, όταν ε, χειραφετούμε τις ε, ανήλικες γυναίκες, αυτό είναι σαν να ε, κόβει τα πόδια στους τρομοκράτες. Και είπαν επίσης ότι μια κοινωνία η οποία επενδύει στη χειραφέτηση των γυναικών τότε θα κυβερνηθεί καλύτερα, θα έχει λιγότερο φανατισμό και όποτε περιορίζονται οι γυναίκες η απασχόλησή τους και η παιδεία τους ε, τότε βρίσκονται σε παρακμή αυτές οι κοινωνίες. Αρχίζει η διαφθορά, και τότε είναι πιο ευάλωτες αυτές οι κοινωνίες στον εξτρεμισμό. Ποιο είναι το μήνυμα ότι η απελευθέρωση των γυναικών όχι μόνο δυναμώνει την κοινωνία αλλά είναι και μια ανάσχεση στον ε, εξτρεμισμό και οπότε έτσι θέλουμε να δούμε πως πολλές φορές θα πρέπει να μην βλέπουμε το, το φαινόμενο τρομοκρατίας και ρισβατικοποίησης μόνο από την πλευρά της ε, ασφάλειας θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι είναι σημαντικός ο ρόλος που παίζουν οι γυναίκες στην ανάσχεση του εξτρεμισμού. Ε, επίσης, ε, πάρα πολύ σημαντικές για την ε, επίλυση των συγκρούσεων και γι' αυτό το 2000 το Συμβούλιο Ασφαλείας με το ψήσμα 1325 ετώνησε χάπου γυναίκες σημαντικές ούτως ώστε να υπάρχει ειρήνευση και να επιληθούν οι συγκρόσεις. Επίσης το Ίδρυμα αναπτυξιακών μελετών απέδειξε ότι οι γυναίκες ενήλικες και ανήλικες μπορούν να βοηθήσουν κάποια προβλήματα σε σχέση με την ειρήνη και την αλλαγή. Είδαμε ότι έγινε με την απαγωγή 300 ανηλίκων γυναικών από την Πόκο Χαράμ στην Ιγυρία και τότε οι γυναίκες πρώτες το κατήγγυλαν αυτό και κάλεσαν να αναλυφθεί μια δράση και χιλιάδες από και μουσουλμάνες στην Ιγυρία φτιάξαν την ομάδα γυναίκες ε, χωρίς ε, τύχη και Επίσης ε, υπήρξε, υπήρξε κάποια συμμαχία στο Πακιστάν κατά του εξτρεμιστικού Αμάνονίσα και στα κράτη-μέλη υπάρχει τέτοια συνειδητοποίηση, υπάρχουν τέτοιες ομάδες γυναικών. Παρά τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά το να λάβουν μέρος οι γυναίκες σε διαπραγματεύσεις για την ειρήνη, μόνο 4% είναι η συμμετοχή των γυναικών σε ειρηνευτικές συμφωνίες. Πολλές φορές οι στρατηγικές κατά της ε, βίας και του εξτρεμισμού παραγνωρίζουν τον ρόλο που μπορεί να λάβουν οι γυναίκες. Και οι εξτρεμιτές ξέρουν ότι οι γυναίκες ε, είναι ένα στοιχείο πολιτισμού στην κοινωνία. Και είδαμε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και πόσο οι συμπαθούντες στο Ισλαμικό κράτος στρέφονται κατά των γυναικών γιατί ξέρουν ότι μπορούν να βοηθήσουν κατά της ζωσοπαστικοποίησης γιατί κάνουν τόσες προσωπικές ε, θυσίες για να προλάβουν την ριζοσπαστικοποίηση. Στο λίγο χρόνο που μου απομένει, να σα πω τώρα για τον ρόλο των σχολείων. Το, η Βρετανική κυβέρνηση πρόσφατα ε, υιοθέτησε ένα νομοθέτημα σε σχέση με το ότι θα πρέπει τα σχολεία να κάνουν κάτι ούτως ώστε να μην ε, στρατολογούν οι τρομοκράτες ε, ανήλικους. Και πρόσφατα στοιχεία κατατείνουν στο ότι ε, σχεδόν οι μισές παραπομπές στην ε, δικαιοσύνη αφορούν ανηλίκους. Και είπαμε ότι πρόκειται για άτομα κάτω από τα 18 και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόβλημα γιατί χρειάζεται να υπάρχει υποστήριξη και πλαισίωση σε πρώιμη φάση της ζωής. Μιλάμε για παιδιά που είναι στο γυμνάσιο και θέλουν να γίνουν ε, ε, μηχανικοί ας πούμε και από τότε ξεκινάνε. Ε, πρώτα πρώτα ξεκινάνε με την αποξένωση από τους φίλους και για τη Λέιλα που ήταν μια τέτοια περίπτωση έλεγε ότι μια παιδεία δυτική δεν πρόκειται να της ασφαλίσει μια θέση στον παράδεισο. Και αυτό το οποίο έπρεπε η Λέιλα να κάνει είναι να ακολουθήσει την Ισλαμική παιδεία. Τι έπαθε η Λέιλα. Το σχολείο είπε τι συμβαίνει στους γονείς. Οι γονείς ανακοφίστηκαν γιατί και αυτοί ήξεραν ότι κάτι συμβαίνει αλλά δεν ξέραν τι να κάνουν. Οπότε παρεπέμφθη η Λέιλα ε, στο σε κάποιο φορέα που λέγεται κανάλι και την βοήθησαν να ξεκαθαρίσει από το μυαλό της τις ακραίες διδαχές του Ισλάμ. Δεν ήταν θέμα αστυνομία, αλλά το σχολείο ήταν ε, ο πρωταγωνιστής του, ώστε να προληφθεί η ριζοπραστικοποίησή της. Θα πρέπει επίσης να κηρυχθούν κάποιες ε, παγκοσμίες αξίες κατά της ε, ακραίας ιδεολογίας, θα πρέπει επομένως να διδαχθούν και οι βασικές αξίες της Βρετανίας, δημοκρατία, κράτος δικαίου, ατομικές ελευθερίες και αμοιβαίος ε, σεβασμός και σεβασμός των διαφορετικών πιστεύω και των ιδιών των άλλων. Και ακριβώς έτσι υπάρχει προστασία. Και ακριβώς όπως λέμε ότι θα πρέπει να, προστατευτούν τα παιδιά από, την γενετήσια... από τον γεννήσιο ακροτηριασμό και την σεξουαλική εκμετάλλευση και θα πρέπει να προστατευτούν και από την ριζοσπαστικοποίηση. Το προσωπικό να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε να υπάρχουν πολιτικές αντίστοιχες. Αλλά υπάρχουν και πολιτικές και για την πληροφορική. Είναι θετικό αυτό που έκανε η κυβέρνηση, ότι αυτή η προσπάθεια ε, νομοθετήθηκε. Προβλέπεται νομοθετικά, οπότε είπαμε ότι έχουμε τώρα ε, εκπαίδευση των ε, μαθητών αλλά και των γονέων για τη ριζοσπαστικοποίηση. Οπότε αναγνωρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο τη σημαντικότητα του προβλήματο. Κάποιοι λένε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι αστυνομικού χαρακτήρα και ότι κανείς κατασκοπεύει τη ζωή του κόσμου και ότι αυτό είναι και η Ισλαμοφοβία. Αλλά όλα αυτά είναι αναλυθεί είναι λάθος. Γιατί έτσι τώρα τα, στα σχολεία ε, υπάρχει συζήτηση, υπάρχει ανοιχτός διάλογος. Και για κάποιους μαθητές μόνο στο σχολείο μπορούν να συζητήσουν αυτές τις ιδέες. Ε, ιδίως όταν ο εξτρεμισμός έχει ήδη φωλιά στην οικογένειά τους. Μα, μας είπε κάποιο παιδί ότι ο πατέρας του ήταν μέλος ε, κάποιας ακραίας το είπε αυτό ένα γόρι και ένα κοριτσάκι. Οι Ισλαμικές ακραίες απόψεις κλπ. Οπότε είπαμε ότι αυτό το σχολείο μπορεί να το καταφέρει, μπορεί να λάβει αυτόν τον ε, ρόλο. Και εν κατακλείδη θέλω να σας πω ότι θα πάρει χρόνο ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή την κατάρτιση των ε, καθηγητών και δασκάλων και είπαμε ότι θα πρέπει να, κατα... να γίνει κατονετή η διαφορά μεταξύ εξτρεμισμού και φυσιολογικών ε, κινήσεων του λειτουργικού του Ισλάμ. θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα παιδιά όσον αφορά τι εξτρεμιστικέ απόψει. Ε, να βοηθήσουν τα παιδιά να μην πέφτουν σε λάθο και να μην ε, αποξενώσουμε του ε, μουσουλμάνου. Πολύ σημαντικά τα σχολεία προστατεύουν τους μαθητές από τη ριζοσβαστικοποίηση κάνουν τα παιδιά ανεφεκτικά σε αυτές τις επιρροές εκθέτουν τους ε, εξτρεμιστές και δίνουν στα παιδιά τον τρόπο να αναλύσουν, να αξιολογήσουν ό,τι διαβάζουν. Εδώ θα το βάλω τελεία και σας ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε για την ε, επιτόπου εμπειρία σας. Your, ε, your, personal and, and, also theoretical. Και δεν είναι μόνο πρακτικά και θεωρητικά ε, και το στρατηγικός ρόλος των γυναικών οπωσδήποτε. Η ΜΚΟ και τα σχολεία ε, που θα πρέπει να συμμετέχουν ε, τα παιδιά, οι δάσκαλοι αλλά και ιδίω οι οικογένειες χωρίς αποκλεισμούς και βεβαίως έχουν ευθύνη και τα μίδια και το διαδίκτυο. Και φαντάζομαι ε, ότι αυτό που λέτε ότι το σχολείο είναι ε, ο μόνος τόπος που μπορούν να ε, προληφθούν αυτά τα φαινόμενα για κάποιους νέους που δεν έχουν άλλη καταφυγή. Δεύτερος ομιλητής μας τώρα είναι, μια στιγμή να το βρω, γιατί κάνω λάθος, είναι ο κύριος Κρίστιανσεν. Έχετε το λόγο παρακαλώ και μετά ερωτήσεις και απαντήσεις ε, όταν θα τελειώσει ο πρώτος γύρος. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω το θέμα μου και πώς η διδασκαλία της ιστορίας μπορεί να προλάβει τη ριζοσπαστικοποίηση. Ας δούμε πρώτα μια παράθεση όταν συναντούν άλλα αφηγήματα και άλλες ιστορίες που αντικρούν ε, αυτά που πιστεύουν κάποιοι, ε, επηρεάζεται και ε, η πληροφόρηση και η συμπεριφορά κάποιου. Και έτσι προάγεται η ανοχή και η ανεκτικότητα. Okay, let's see. Okay. So... Λοιπόν, Πώς μπορεί η ιστορία, η διδασκαλία της ιστορίας να συνεισφέρει ε, στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Γι' αυτό θα σας μιλήσω. Εκπροσωπώ εδώ την Euroclio που είναι ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Διασκόντων Ιστορίας. Ε, Έχουμε 48 ανεξάρτητα σωματεία που είναι μέλη μας ε, που ε, τα μέλη διδάσκουν ιστορία και αγωγή του πολίτου από 47 χώρες και στις 17 Μαρτίου φέτος οι Υπουργοί Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωση συναντήθηκαν στο Παρίσι και συμφώνησαν για μια διακήρυξη που καλεί ε, σε δράση ή μεταξύ άλλων να ενισχύσουν το ρόλο της εκπαίδευσης, την πρόθεση ε, της αγωγής του πολίτη και τις κοινέ αξίες ελευθερίας, ανεκτικότητας και μη διάκρισης, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και βοηθώντας τους νέους να αποκτήσουν ευθύνε και να έχουν ανοιχτό πνεύμα και να είναι ενεργά και πλήρη μέλη μιας κοινωνίας ε, με πολυμορφία και χωρίς αποκλεισμούς κατά τη διάρκεια ε, της ε, διάσκεψης στο Χέλσιγκορ της Δανίας, λίγες εβδομάδες μετά, 157 ιστορικοί και καθηγητές αγωγής πολίτου από 40 ε, χώρες εργάστηκαν επί αυτού του θέματος και κατέληξαν στη διακήρυξη του Χέλσιγκορ μετά τη διακήρυξη των Παρισίων. Και το βασικό μήνυμα ήταν το εξής. Είναι σημαντική η έκκληση ε, της ε, διάσκεψης των Παρισίων και της διακήρυξης και η ιστορία μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται η ιστορία. Και επανέρχομαι στη δική μας αποστολή. Το Ευρωκλειό έχει στόχο να ε, διδάσκει την ιστορία και να φτιάχνει πολίτες υπεύθυνου καινοτόμου με κρίσιμη σκέψη, κριτική μάλλον σκέψη και αυτό θα βοηθήσει για την ενίσχυση του αλληλοσεβασμού, της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Τι σημαίνει υπεύθυνη διδασκαλία της ιστορίας. Θα πρέπει να βοηθούμε τους μαθητές να καταλαβαίνουν ότι η ιστορία είναι ερμηνεία των ιστορικών πηγών, θα πρέπει να τις διασταυρώνουμε, να τις συγκρίνουμε έτσι ώστε να έχουμε επιχειρήματα για να απαντούμε σε ερωτήσεις. Με κριτικό βλέμμα. Και πάντα η ιστορία είναι περίπλοκη. Κάθε απάντηση οδηγεί σε νέες ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλά επίπεδα και πολλές σχέσεις. Είναι περίπλοκο αυτό το θέμα και το αφήγημα πάντα είναι ένα εργαλείο επιλεκτικό. Και τέλος, η ιστορία βασίζεται σε αξίες. Απαντά σε ε, σημερινές συμπεριφορές και ε, σε μενά θέματα. Άρα λοιπόν μια υπεύθυνη δασκαλία της ιστορίας ε, είναι κάτι που εξετάζει πολλούς τομείς και διεπιστημονικά. Για να γίνει αυτό όμως στα σχολεία ε, σε σχέση με την δημόσια ιστορία, την ακαδημαϊκή έρευνα και την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αρνητικά. Υπάρχει και πολιτική χρήση και κατάχρηση της ιστορίας. Ε, για να γίνει με το σωστό τρόπο η διδασκαλία θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές για να μάθουν να μαθαίνουν και να αναπτύξουν αυτή την ιστορική συνείδηση. Βάσει λοιπόν των παρατηρήσεων και των πολιτικών μας, οι συμμετέχοντες ε, στην ε, διάσκεψη του Χέλσιγκορ είπαν τα εξής και έθεσαν στόχους για την διακήρυξη του Παρισιού έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε για τη δασκαλία της ιστορίας. Για να αναλάβουμε τη δράση λοιπόν που ζητεί η διακήρυξη του Παρισιού θα πρέπει να αναπτύξουμε νέα εκπαιδευτικά εργαλεία και πηγές, να υποστηρίξουμε τα ρυθμίσεις των προγραμμάτων των σημερινών ε, και του τρόπου εξέτασης για να υπάρξει ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Πώς θα γίνουν όμως όλα αυτά. Πρέπει στο κέντρο να είναι ο μαθητής σε ό,τι αφορά την ταυτότητα, την ε, διαμόρφωση γνώμης και την ενημέρωση σε μια ψηφιακή εποχή. Επίσης, χρειάζεται μια παιδαγωγική συνεργασίας και ποιότητας ε, και μια διδασκαλία της ιστορίας που να αντανακλά την πολυμορφία. Ποια είναι τα μηνύματα λοιπόν είναι μηνύματα που βασίστηκαν στην παρακολούθηση της σημερινής διδασκαλίας της ευρωπαϊκής ιστορίας. Σε κάποιες χώρες ε, βλέπετε μαθήματα ιστορίας που, και βιβλία και σχολικά εγχειρίδια που περιλαμβάνουν έννοιες όπως είναι η κριτική σκέψη, η εκπαίδευση των πολιτών, δημοκρατία, ανεκτικότητα, πολυμορφία, διαφορετικότητα. Αν δείτε όμως τις τελευταίες σελίδες ε, των εγχειριδίων, συχνά ε, και των προγραμμάτων εκπαίδευσης θα δείτε ένα στάνταρ τρόπο εξέτασης ε, αλλά τι μαθαίνουμε, τι διδάσκουμε. Συνήθως μιλάμε για πολέμους, για πολιτική και για άντρες Άρα υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στους στόχους και τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται και εξετάζεται τελικά το μάθημα της ιστορίας. Για ποιο λόγο Έχω έρθει εγώ εδώ σήμερα ως δανός καθηγητής ιστορίας. Ε, είναι τα βιβλία μας και το σύστημα με τον οποίο, το οποίο εκπαιδεύουμε. Ε, στην εισαγωγή μας του βιβλίου της ιστορίας θα δείτε τα ίδια στοιχεία που έχουμε σε όλη την Ευρώπη. Κριτική σκέψη, ε, παιδαγώγηση πολιτών, δημοκρατία, ανοχή και πολυμορφία. Όταν φτάσουμε όμως στις τελικές εξετάσεις θα διαβάσετε το εξής αποφασίζει το κάθε σχολείο ε, τι εξέταση θα κάνει ε, με βάση ε, κάποιο πρόγραμμα στο οποίο έχουν συμφωνήσει στο μάθημα καθηγητές και τάξη με βάση τους στόχους που έβαλαν στην αρχή και συζητούν οι μαθητές, παρουσιάζουν και συμμετέχουν. Στο γυμνάσιο ή στο λύκειο στη Δανία υπάρχει διάλογος του παρόντος με το παρελθόν. Πάντα αυτή είναι η αφετηρία μας στην ιστορία. Ε, πολιτισμικές συναντήσεις, ταυτότητες, μετανάστευση, δημοκρατία, μέσα Ανατολή, ε, μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Είναι ε, μαθήματα ε, και αντικείμενα που διδάσκεται ο Δανός στο γυμνάσιο. Άρα γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο να αντιστοιχηθούν οι στόχοι με ε, την εξέταση και το τι ζητάμε από το μαθητή να μάθει στο τέλος. Η βασική ιδέα λοιπόν, η κεντρική ιδέα είναι ως εξή του δανεικού συστήματος. Οι εξετάσεις μας θα πρέπει να ε, είναι αντανάκλαση της καθημερινής ζωής μέσα στην τάξη. Και η καθημερινή ζωή μέσα στην τάξη θα πρέπει με τη σειρά της να είναι αντανάκλαση της ζωής της καθημερινής. Το 2009 ε, ο τότε Υπουργό Παιδείας είναι νυν Υπουργό ε, Πολιτισμού στη Δανία. If we put together... Λοιπόν, εάν ε, συνδυάσουμε λοιπόν τη διακήρυξη των Παρισίων και όσα λέγουν οι Δανείοι μαθητές και τα συγκρίνουμε, τι θα διαπιστώσουμε. And Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν το δανεικό παράδειγμα και την πρακτική ευρωκλειό καταλήγει. Η διδασκαλία της ιστορίας μπορεί με σημαντικό τρόπο να συνεισφέρει στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. On Στη βάση λοιπόν αυτής της παρουσίασης η Ευρωκλειό έχει προβήσει συστάσεις για την Επιτροπή σας προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, διευκολύνει το Erasmus Plus έτσι ώστε να μπορούν ε, να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν οι επαγγελματίες. Ε, και το Ορίζον 2000 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτός από τον Erasmus ε, Plus και ε, κάποια άλλα εργαλεία να ενισχυθεί η συνεργασία. Επίσης να ενισχυθεί ο της ευρωπαϊκής ιστορίας ως ένας χώρος ιστορικού διαλόγου για τη μετανάστευση και την ε, διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει μια πλατφόρμα για το ρόλο της εκπαίδευσης σε αντιπαράθεση με την ασφάλεια συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχουν τα πλαίσια όπως είναι η αγωγή του δημοκρατικού πολίτου, η αγωγή στα ανθρώπινα δικαιώματα και η αγωγή για την παγκόσμια ηθαγένεια. Και τέλος, θα πρέπει να σκεφτείτε ότι οι επενδύσεις στην παιδεία είναι μακράς πνοής και δεν έχουν ταχεία απόδοση. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Σαφέστατη παρουσίαση και πολύ ενδιαφέρουσα. Σίγουρα θα βοηθήσουν όλες αυτές οι απόψεις ε, την Επιτροπή μας και θα εμπλουτίσει τις εκθέσεις της. Θα Έχουμε τώρα ένα γύρο ερωταπαντήσεων. Ο κύριος Σιβέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και για την οργάνωση της δημόσιας ακρόσης ε, με το συγκεκριμένο αυτό θέμα που είναι εξαιρετικά επίκαιρο και χαίρομαι ιδιαίτερος που προσκαλέσαμε ε, τόσους, τόσο σημαντικούς και διακεκριμένους ε, εμπειρογνώμονες στην σημερινή μας δημόσια κρόση. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Σαρακάν, της Διευθύντριας του Φορέα Inspire, που στήριξε την παρουσίασή της στις ε, προσωπικές της εμπειρίες και μας έδειξε πως ε, μερικοί δίνουν μάχη για το δημοκρατικό διάλογο πώς δίνουν μάχη για μια καλύτερη κοινωνία που θα επιτρέπει τέτοιο δημοκρατικό διάλογο. Βέβαια, θα πρέπει να φροντίσουμε να υιοθετήσουμε μια συνολική προσέγγιση. Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να λάβει μέρος στη συζήτηση αυτή η Εκκλησία το ίδιο και άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα πρέπει να εμπλακούν στην προσπάθεια αυτή. κυρία Χάν μας μίλησε για το ρόλο των γυναικών. Ένα αξιοσημείωτο θέμα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερος, γιατί ο ρόλος των γυναικών πολύ συχνά παραμελείται και ειδικά στο Ισλάμ, ενώ οι γυναίκες μπορούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην παιδεία και την ανατροφή των παιδιών. Όταν βλέπουμε όμως το ρόλο των γυναικών στην παιδεία, διαρωτόμαστε και οι άντρες τι κάνουν στο θέμα της παιδείας. Στη δική μου πατρίδα έχουμε άλλο φαινόμενο. Το εκπαιδευτικό σύστημα γυναικοκρατείται. Η πλειοψηφία των διδασκόντων του διδακτικού προσωπικού είναι γυναίκες. Πώς θα, εντάξουμε λοιπόν και τους άνδρες σε αυτή τη διαδικασία στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις θέσεις των διδασκάλων και καθηγητών. Επίσης, η πρωτοβουλία Κλείο μας παρουσίασε ο κύριος Κρίστενσεν διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο τις τελευταίες δεκαετίες για να απεθνικοποιήσουμε τα σχολικά προγράμματα ή τα προγράμματα σπουδών. Ναι. Και όταν το 1990 άρχισαν να, δημιουργούνται νέες ε, χώρες μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, διαμόρφωσαν τα προγράμματα σπουδών τους, αλλά αυτά δεν ανταποκρινόταν τότε στην πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλουμε στην ανέβρεση μιας λύσης για να δημιουργήσουμε ένα κλίμα και μια ατμόσφαιρα πρόσφορε για διάλογο διαπολιτισμικό. Τώρα μας απασχολεί η προσφυγική κρίση. Δεν θέλουμε να αναπτυχθούν διάφορες κοινωνίες ή κατακαιρματισμένες κοινωνίες και θα χρειαστούμε μηχανισμούς και εργαλεία για να αποφύγουμε τέτοιο κατακαιρματισμό. Ευχαριστώ. Σε λίγο πρέπει να φύγω. Έχω υποχρεώσει στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θέλω να προλάβω να ακούσω και τις απαντήσεις. Κύριε Κρίστιανσεν, είπατε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η οίκη της ευρωπαϊκής ιστορίας για να ενισχυθεί, να διευκολυνθεί ο ιστορικός διάλογος για τη μετανάστευση και ούτε καθεξής. Μήπως έτσι όμως ε, δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος ε, της προσέγγισης. Δεν νομίζω ότι θα έχετε τη συντριπτική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Πώς λοιπόν θα συμβάλλουμε ώστε να ληφθεί υπόψη η ανησυχία τους. Ας ακούσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους που έχουν απορίες, σχόλιο. Ο κύριος Κρασνοντέμψκι. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις και οι διεμπειρογνώμονες μας είπαν πολύ σημαντικά πράγματα. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο ρόλος των γυναικών. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό θέμα κέρυες σημασίας. Γιατί μία από τις μεγάλες διαφορές που έχουμε είναι η σημασία που δίνουμε στο ρόλο της γυναίκας. Εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Είπατε στην ομιλία σας, κυρία Χάν, ότι Υπάρχει μια γραμμή που είναι δύσκολο να την ε, χαράξουμε στην πραγματικότητα μεταξύ του εξτρεμισμού αφενός και της αποδοχής των πολιτισμικών διαφορών αφετέρου και των πολιτικών συμπεριφορών επίσης. Θα πρέπει λοιπόν με πολύ προσοχή να προσδιορίσουμε ποια είναι μια ριζοσπαστική άποψη που είναι απαράδεκτη και πότε έχουμε δικαίωμα παρέμβασης ή επέμβασης. Γιατί όταν ακούμε τη λέξη παρέμβαση, αντιδρούμε. Είπατε ε, ότι ένας από τους γονείς ήταν πολύ συντηρητικός. Και εγώ το ίδιο. Θεωρώ ότι είμαι συντηρητικός ε, πατέρας και δεν θα ήθελα να επεμβαίνει στο έργο μου ε, το σχολείο. Και μάλιστα ως μετανάστης και προσκεκλημένος Πολωνός καθηγητής δίδαξε σε Γερμανικό Πανεπιστήμιο. Και μερικές φορές οι γερμανοί καθηγητές ε, δεν κατάλαβαν πόσο σημαντικό ήταν για μένα να ε, μεταλαμπαδεύσω αυτή την πολωνική κουλτούρα στην κόρη μου. Γιατί θεωρούν ότι είμαστε εμείς πιο συντηρητικοί ε, από θρησκευτική απόψεις. Οπότε πρέπει να βρούμε αυτή την διαχωριστική γραμμή που είναι δύσκολο να βρεθεί μερικές φορές. Μετά ο κύριος Κρίστενσεν μας είπατε πώς θα πρέπει να διδάσκουμε την ιστορία. Βέβαια, η διδασκαλία της ιστορίας έχει και άλλες λειτουργίες. Την προάσπιση της εθνικής ταυτότητας, την ε, μεταβίβαση της ε, ταυτότητας, της ιστορικής ε, μνήμης από, από τη μια γενιά στην άλλη. επίσης διδασκόμαστε από τις αξίες του παρελθόντος και μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι ο τρόπος διδασκαλής της ιστορίας δεν είναι μόνο το φάρμακο κατά του εξτρεμισμού και του, της ριζοσπαστικοποίησης, γιατί ο ορισμός της ριζοσπαστικοποίησης είναι η βία. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Η, η ροπή προς ε, τα τρομοκρατικά κινήματα. Και αυτή η τέχνη της δασκαλίας ε, της ιστορίας είναι σημαντική. Αλλά θεωρείται ότι είναι λάθος ως ε, δανός ιστορικός ε, να είστε και δανός πατριώτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι όντας κάποιος πατριώτης θα είναι αρνητικός απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους. Αλλά μπορεί κανείς επιβεβαιώντας και τετρανώντας την ταυτότητά του να λαμβάνει έτσι μια, ιστορική, μια θέση απέναντι στην ιστορία. Αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να δείξουμε ανοχή και στους υπόλοιπους. Ή κάποιος που θέλει να προβάλλει την θρησκευτική του ταυτότητα ή την εθνική του ταυτότητα, δεν είναι το ίδιο με έναν εξτρεμιστή, έναν ριζοσπάστη που είναι δημόσιος κίνδυνος. Προσοχή λοιπόν, ακόμη και στην ιστορία, δεν θα πρέπει τη γραμμή να τη χαράζουμε σε λάθος σημείο. Ε, Τρούπελ. Η κυρία Τρούπελ, σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα επίσης να σταθώ σε αυτά που είπε η, η, η κυρία Κάμπτη, δηλαδή αποστερεί τα δικαιώματα της γυναίκας στο Ισλαμισμό. Οπότε θα πρέπει επομένω ε, να ανασχέσουν την ζωσπαστικοποίηση γυναίκες. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα. Και επίσης Υπάρχουν ένα σωρό στοιχεία που έχουμε στα χέρια μα, αλλά και προγράμματα. Και έτσι μπορούμε να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Επίση, δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Σαρακα, ότι οι μουσουλμανοί είναι ένα πόσο τμήμα των κοινωνιών όπου ζουν. Και δεν θα πρέπει να του βλέπουμε ε, σαν κάποιους ε, που είναι εκτό κοινωνία. Γιατί αυτό είναι ακριβώ και το πρόβλημα με του νέου, ότι δεν αισθάνονται μέρος της κοινωνίας όπου ζουν. Επομένως ε, σε αυτό το μέτωπο να δουλέψουμε σκληρά. Και τώρα το τελευταίο είπα την κύριε Τέρσκι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της θεμελιώδους αξίας της ελευθερίας του πιστεύει και το να αποκλίνει κανείς προς εξτρεμιστικές απόψεις. Γιατί ε, δεν είναι μόνο η βία, είναι και η έκφραση του μίσους και είναι και το να αποστερεί κανείς από άλλον την ε, αξιοπρέπειά του. Οπότε θα πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση μεταξύ της ελευθερίας ε, της θρησκευτική και την άλλη μεριά του να παρασύρεται κανείς από εξτρεμισμό και να αποστερεί από άλλους τα δικαιώματά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτά τα οποία είπατε λέει η Πρόεδρος. Αυτά τα σχόλια σε σχέση με τόσο είπε δουλεύετε και με διάφορους φορείς και μη κυβερνητικέ οργανώσεις και επίσης είναι σημαντικός και ο διαθρησκευτικός ε, διάλογος. Εκεί να συζητείτε το πρόβλημα. Γιατί ε, νομίζουμε ότι όταν κανείς συζητά στα πλαίσια των περισσότερων θρησκειών, τότε υπάρχει περισσότερη λοκατανόηση. Και η ιστορική διάσταση ήταν πολύ σημαντική, κύριε, κύριε καθηγητά, που είπατε ότι θα πρέπει να βοηθούμε στην κατανάλωση, στην κατανόηση. Και να δούμε πώς θα μπολιάσουμε στο πρόγραμμα διδασκαλίας την ανοίξη της διαφορετικότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θέλετε να απαντήσετε, έχετε το λόγο. Κρίστενσον. Όχι. Κύριε Χάν, μία ερώτηση νομίζω απευθύνθηκε απευθεία σε μένα. Υπάρχει διαφορά, όπως είπαν οι συνάδελφοι, μεταξύ της κουλτούρας και του σεβασμού της της θρησκευτικής και πολιτισμικής πολυμορφίας, ε, του δικαιώματος ανεξαθρησκείας, γιατί αυτό συνιστά το μεγαλείο της Ευρώπης ε, και αυτό μας διαχωρίζει από τους δικτάτορες, τους τυράννους. Αυτό μας ε, κάνει μια μεγαλειώδη δημοκρατία, ακριβώς η ικανότητά μας να σεβόμαστε τις διαφορές. Και οι μειονότητες να μπορούν να δίνονται διαφορετικά, να τρώνε διαφορετικά, να, έχουν, να πρεσβεύουν διαφορετικά πράγματα, να έχουν διαφορετική θρησκεία. Αυτή η πολυμορφία, η διαφορετικότητα είναι θετικό στοιχείο και όχι αρνητικό και η ιδέα μου για τον εξτρεμισμό. Και υπάρχει και θέμα τι εννοούμε, πώς ορίζουμε τον εξτρεμισμό. Γιατί φαντάζομαι κάθε χώρα ορίζει διαφορετικά τον εξτρεμισμό. Και ε, ακόμη και για τον ορισμό της τρομοκρατίας καθυστερήσαμε πολύ για να καταλήξουμε σε ένα κοινό. Τώρα συμφωνήσαμε. Αλλά το να ορίσουμε τον εξτρεμισμό είναι ακόμη πιο δύσκολο από το να ορίσουμε την τρομοκρατία όπως καταφέραμε μετά από πολύ καιρό. Η Βρετανική κυβέρνηση θεωρεί ως ενεργό ή προφορική ε, αντίσταση στις θεμελιώδεις αρχές. Αυτό θεωρεί εξτρεμισμό η Βρετανική κυβέρνηση. Τι είναι όμως οι θεμελιώδεις αρχές. Είναι δύσκολο να ορίσουμε λοιπόν τον εξτρεμισμό. Εγώ θεωρώ ότι ο εξτρεμισμός είναι η υποδάβληση του μίσους, της βίας, η εξύμνηση του μίσους, η προσπάθεια να αποστερήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα συνανθρώπων μας, η ανισότητα μεταξύ των φίλων. Εγώ είμαι φεμινίστρια και αν κάποιος ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες δεν είναι ίσες ε, με τους άνδρες, ε, θεωρείται κανείς εξτρεμιστής με τις αξίες του 21ου αιώνα που πρεσβεύουν την ισότητα. Όλοι δίνουμε μάχη και ίσως μετά από μερικά χρόνια κάποιος που δεν θεωρεί ότι τα δύο φύλλα είναι ίσα θα θεωρείται εξτρεμιστής. Και για να, να προλάβουμε την ριζοσπαστικοποίηση θα πρέπει να δούμε ποιες ιδεολογίες εξυμνούν και προωθούν ε, το μίσο ή, χρη... ή χρησιμοποιούν τη ρητορική του μίσου. Αυτό το κάνουν και εξτρεμιστικέ ομάδε, αλλά και ακροδεξιέ ομάδε, για παράδειγμα. Και μερικοί το πάνε ακόμη πιο μακριά. Περνάνε από τα λόγια στα έργα, στη χρήση τη βία. Και αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αλλά αυτό είναι τελείω διαφορετικό από το σεβασμό τη πολιτισμική πολυμορφία. Γιατί αυτό το νόημα έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η χρησιμοποιουν τη ρητορικη του μίσου. αυτο το κανουν και εξτρεμιστικε ομάδε, αλλα και ακροδεξιέ ομάδε, για παραδειγμα και μερικοι το πανε ακομη πιο μακρια περνανε απο τα λογια λοιπόν, στα εργα στη χρηση τη βία. και αυτο ειναι κατι πολυ διαφορετικο αλλα αυτο ειναι τελείω διαφορετικο απο το σεβασμο τη πολιτισμικη πολυμορφιας γιατι αυτο το νοημα σημαντική. Επίσης, ε, μιλήσατε για τις υπόλοιπες ε, θρησκείες και δοξασίες. Ε, εγώ συνεργάζομαι με ομάδες χριστιανών, Εβραίων, αλλά και με ομάδες με λαϊκό προσανατολισμό ανθρωπιστικό. Η συνεργασία με ομάδες, με κοινότητες Εβραίων είναι πολύ σημαντικές, γιατί το Ισραηλοπαριστηλιακό πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα όταν έχουμε δολοφονίες εκεί, έχουμε μια έξαρση του αντισημιτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο με το που ε, ενισχύεται η βία στην, στην Παλαιστίνη. Και το αντίστροφο επίσης έχουμε διαπιστώσει. Όταν έχουμε μια τρομοκρατική επίθεση, έχουμε έξαρση του αντιμουσουλμανισμού. Είχαμε το 2012 ε, τέτοιες τρομοκρατικές ε, επιθέσεις και αντίστοιχη έξαρση του αντιμουσουλμανισμού. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαστούμε με τις διάφορες κοινότητες, ε, τις θρησκευτικέ και τις λαϊκές. Και όλοι από κοινού να συμφωνήσουμε στις αρχές της δημοκρατίας, της λαϊκοσμικότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί πολλές τέτοιες ομάδες ε, της κοινωνίας των πολιτών εφορούνται από τέτοιες αρχές. Ευχαριστώ κύριο Κρίστενσεν. Ευχαριστώ. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να τονίσω κάποια στοιχεία για το πώς διδάσκεται η ιστορία σε μια κοινωνία. Τι πιστεύω εγώ και τι πιστεύει και η δική μας Ένωση. Είναι βασική μας ευθύνη να απαντάμε στις προκλήσεις και στις εμπειρίες που έχουν οι σημερινοί μαθητές και φοιτητές ε, πριν καν διαμορφώσουν ιστορική συνείδηση. Και έτσι χρειάζονται και τα απαραίτητα εργαλεία και εκπαίδευση για τους στόχους που έχουμε θέσει. Και νομίζω αυτό είναι παντού σε όλα τα προγράμματα σπουδών, η διδακτέα ύλη, σε όλη την Ευρώπη. Ανοχή, ε, ενεργός πολίτης, συμμετοχή, ε, πολυμορφία κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διδάσκοντες στην ιστορία έχουν τα έργα λία εκείνα ε, που εμφορούνται από μια πολιτική ατζέντα. Καθόλου. Εμείς δεν διαβιβάζουμε ε, μία ε, ιστορική αλήθεια, μία πολιτική αλήθεια. Δεν είμαστε κοινωνιολόγοι, δεν είμαστε κοινωνικοί λειτουργοί. Και δεν βαθμολογούμε τους ε, μαθητές μας με βάση το επίπεδο ανοχής και ανεκτικότητας που επιδεικνύουν. Είμαστε επαγγελματίες. Αυτό που θέλουμε είναι οι φοιτητές και οι μαθητές μας να είναι προετοιμασμένοι να μπουν σωστά στην ενήλικη ζωή τους. Και Ξέρουμε ότι αυτό δεν περνάει μέσα από τη δασκαλία της ιστορίας και μόνο, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Να έχουν εκπαιδευτεί στην κριτική σκέψη. Να βλέπουν ένα θέμα από πολλά πρίσματα και οπτικές γωνίες και να μπορούν να είναι σε ένα μόνιμο και διαρκή διάλογο του παρόντος με το παρελθόν μέσα στο μυαλό τους. Και έρχομαι στις ερωτήσεις που μου κάνατε. Για τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Όχι. Δεν είναι καθόλου προσέγγιση ε, που έχει επιβληθεί από την κορυφή προς τη βάση, από πάνω προς τα κάτω. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι πώς να το πω, να υπάρχει ένας φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μπορεί να κάνει μαθήματα και εντός του μουσείου και στα κράτη-μέλη και να διαδίδονται ε, βέλτιες πρακτικές ε, την καταπολέμηση των αποκλεισμών και να συζητούμε. Και δεν θα καταλήγουμε στη μία την απόλυτη αλήθεια ή δυνατόν, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να εξετάζουμε πώς το βλέπουν οι διάφορες χώρες και πώς το χειρίζονται. Και έρχομαι τώρα στην άλλη ερώτηση. Σήμερα το θέμα μας είναι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Και γι' αυτό επικεντρωθήκαμε ακριβώς σε αυτά τα σημεία και τη διακήρυξη των Παρισίων που ζητεί δράση. Βεβαίως, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ιστορίας. Ε, φυσικά η βάση είναι η εθνική ιστορία. Πάντα θα διδάσκεται αυτή. Και όλοι θέλουμε να αισθανόμαστε γιατί ζούμε σε μια πολύ καλή χώρα. Και η ιστορική εκπαίδευση και αυτό θα πρέπει να το υποστηρίζει, να μαθαίνει ο καθένα την ιστορία του. Αλλά τι βλέπουμε, καμιά φορά κατά τη γνώμη μου, το παρακάνουμε στον ενθουσιασμό και ξεχνάμε να συμπεριλάβουμε και τις μειονότητές μας σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε εθνικό αφήγημα. Η δική μου ένωση επιμένει πάρα πολύ σε αυτό και μας ενδιαφέρει και στα διεθνή εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Βεβαίως χρειάζεται μια ισορροπία οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ. Story of hm? Είναι, δεν είναι η ιστορία των ιστοριών. Είναι πολλές ιστορίες που κάνουν την ιστορία. Μισό λεπτό. Ναι, δύο, δύο λέξεις μόνο θα πω. Βλόγα ε, Λοιπόν, ήθελα να πω για το ρόλο των ε, διδασκόντων και ο ρόλος της ιστορίας δεν είναι μόνο να ζητήσει την ιστορική αλήθεια, αλλά και να δείξει στους νέους ότι τι σημαίνει και τι έχει ιστορική σημασία και τι δεν έχει. Τι ήταν σωστό και τι λάθος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε στους νέους μας την αίσθηση του σημαντικού, του ηθικού και ε, του εσφαλμένου. Κυρία Χάν, ο πολιτισμός μας δεν επικεντρωνόταν σε αυτό, στην, στην ισότητα ανδρών και γυναικών στο παρελθόν. Αν είστε όμως στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν τίθεται κανένα δίλημα. Φυσικά και υπάρχει ισότητα των φίλων. και θα πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό. Αυτό άλλωστε το έχουμε ήδη πετύχει. Είναι μια κατάκτηση διαμέσου της ιστορίας. Και πιστεύω πραγματικά ότι και άλλοι πολιτισμοί θα πρέπει να το υιοθετήσουν και θα το υιοθετήσουν και άλλες θρησκείες. Ε, παρατήρηση ή ερώτηση. Περισσότερο. Μια παρατήρηση παρά ερώτηση, λέει η Πρόεδρος. Ωραία, τώρα Μπορεί τωρα μπορουμε να συνεχίσουμε επομένως και τώρα δώσουμε το ε, λόγο στον κύριο Ντεμομπριάλ. Και αυτός έχει 15 λεπτά και εκατόπιν ο κύριος ε, Μπέργκερ από την ΟΝΕΣΚΟ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι, πώς ε, θα προλάβουμε το πολιτισμικό και εδαφικό ρήγμα και το κατακαιρματισμό. Ξέρω ότι δεν είναι ανώδυνε οι λέξει που χρησιμοποιώ, γιατί οι κατάσταση στην Ευρώπη και στη Γαλλία είναι πολύ σοβαρέ, πολύ πιο σοβαρέ από ό,τι μερικοί θέλουν να πιστεύουν ή από ό,τι μερικοί ισχυρίζονται. Η Ευρώπη γενικώ και η Γαλλία ειδικώ αντιμετωπίζουν εδώ και μία διετία περίπου ένα τελείω πρωτόγνωρο φαινόμενο. Ένα τμήμα τη νεολαία μα έχει γίνει το πεζικό ενό πολέμου που γίνεται στην επικράτειά μα στο όνομα μια θρησκεία, ε, προκειμένου του ριζοσπαστικού συνειδητικού Ισλάμ. Ισλάμ. Μάλιστα, η καλπάζουσα αύξηση του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης του Ισλάμ στην Ευρώπη εκφράζεται και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το εύρο, οι διαστάσεις και η σοβαρότητα αυτού του κοινοτιστικού ρήγματος στη Γαλλία φαίνεται και στο εκπαιδευτικό σύστημα και μας δείχνει την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και την οποία θα ξεπεράσουμε όταν σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε μπροστά στι καταστροφικέ συνέπειε που εξηγούνται κυρίω από το γεγονό ότι τα 60 χρόνια ειρήνης που ολοκληρώνουν μα οδήγησαν στο να είμαστε πολύ λιγότερο προσεκτικοί και να έχουμε χαλαρώσει υπερβολικά. Θα σα ε, εξηγήσω εν συντομία πώς ε, αυτός ο κοινοτισμό ε, διακυβεύει και επηρεάζει το εκπαιδευτικό σύστημα και θα σας προτείνω κάποιες λύσεις. Αυτή η έξαρση λοιπόν της κοινοτικής εισπύρωσης, της κοινοτιστικής εισπύρωσης στην Γαλλία φαίνεται από διάφορα επεισόδια και περιστατικά που παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ιανουαρίου του 2015 είχαμε έντονες εντάσεις στα περισσότερα σχολεία της Γαλλίας. Βέβαια, πολλοί πολιτικοί προσπάθησαν να υποβιβάσουν το φαινόμενο και ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας μίλησε για 200 περίπου περιστατικά τέτοια επεισόδια. Ενώ φάνηκε από πολλά στοιχεία ότι πάνω από 200 περιστατικά είχαμε σε κάθε διαμέρισμα. Έχουμε 100 διαμερίσματα στη Γαλλία. Και συγκεκριμένα τα περιστατικά αυτά ε, είτε αναφέρονταν σε ε, ομιλίες που δικαιολογούσαν την πράξη αυτή. Μερικοί ε, καταδίκαζαν τη σοβαρότητα, ε, γιατί ήταν ε, πρόκειτο για δολοφονίες, αλλά τη σχετικοποιούσαν επικαλούμενη την προκλητικότητα των σκητσογράφων εις βάρος του Ισλάμ και του προφήτη. Επίσης, σε όλα τα γαλλικά διαμερίσματα, ούτε σε ένα διαμέρισμα της υπαίθρου δεν είχαμε ηρεμία. Όλοι, σε όλες τα διαμερίσματα είχαμε διαταραχή κατά την τήρηση του ενός λεπτού σιγή. Είχαμε διάφορα περιστατικά, για παράδειγμα διακοπή του λεπτού σιγής, μερικοί μαθητές άρχισαν να τραγουδούν τον αλγερινό εθνικό ύμνο, οι άλλοι να κραυγάζουν Αλάχ Ακμπαρ, στη διάρκεια αυτής της στήριξη του λεπτού σιγής για τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Πολλά τέτοια περιστατικά λοιπόν παντού στη Γαλλία. Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στις 24 Σεπτεμβρίου, 24 Σεπτεμβρίου δηλαδή στην γιορτή του Αίδαλ Κεμπίρ σε πολλά σχολεία της Γαλλίας διαπιστώσαμε απουσία που έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ και μαθητών και καθηγητών. Και μάλιστα στην ΙΜ, σε μια μικρή πόλη της Νότιας Γαλλίας, ε, σε ένας καθηγητής επαγγελματικού λυκείου μου είπε ότι 70 Μαθητέ από του 500 ήταν παρόντε, δηλαδή 430 μαθητέ απουσίαζαν, έκανα κοπάνα και 40 καθηγητές από τους 70 έδωσαν το παρόν εκείνη τη μέρα. Έχουμε λοιπόν τέτοια περιστατικά στο σχολικό σύστημα που ουσιαστικά αντανακλούν άλλα ε, περιστατικά και συμβάντα στο σύνολο της κοινωνία. Για παράδειγμα, όταν ε, έχουμε ποδοσφαιρικούς αγώνε με ομάδε του Μαγκρέμπ ή το Σαββατοκύριακο που έχουμε γάμους ε, στις ε, κοινότητες αυτές, οι τοπικές ε, αρχές αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις ή σε χαρακτηριστικές γιορτές, όπως είναι η Εθνική Εορτή. Για παράδειγμα, εδώ και μερικά χρόνια έχει γίνει παράδοση κάθε 14 Ιουλίου, την Εθνική Εορτή της Γαλλίας, έχουμε παραδόσεις βίας, βίων φαινομένων, έκτροπα, πυρπολούνται αυτοκίνητα. Και στις 14 Ιουλίου πέρυσι για πρώτη φορά είχαμε τέτοιες διαστάσεις και τέτοια διάρκεια ε, της βίας. 17 αστυνομικά τμήματα υπέστησαν επιθέσεις και μάλιστα σε μερικά αστυνομικά τμήματα αντικαταστάθηκαν οι γαλλικές σημαίες από τις ε, σημαίες της Αλγερίας. Τέτοια φαινόμενα πλήττουν ε, τη Γαλλία και μάλιστα έχουν συγκεντρωθεί πολλά τέτοια στοιχεία από τις μυστικές αρχές της Γαλλίας. Βέβαια δεν είναι απλές προκλήσεις που γίνονται κάθε φορά. Πολύ συχνά έχουμε καθηγητές και μάλιστα καθηγητές των μαθημάτων γεωργίας και ιστορίας που δεν τολμούν να διδάξουν κάποια ιστορικά επεισόδια γιατί και μόνο που αναφέρονται σε κάποια εδάφη, σε ιστορικές περιόδους είναι αρκετά για να δώσουν λαβή σε φασαρή στην τάξη και έκτροπα που είναι αδύνατο να τα διαχειριστούν. Λιγότερο σημαντικό, αλλά για κάποιους καθηγητές βιολογίας, ε, χημίας και τέτοιων μαθημάτων επίσης υπάρχουν προβλήματα στην διδασκαλία. Αυτές λοιπόν ε, οι πληγές που αφήνει ο κοινοτισμός, αυτή η κοινοτική συσπήρωση ε, είναι τεράστιες και δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για τη στρατολόγηση του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Αρισυχητικά τα νούμερα στη Γαλλία. Χθε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών μίλησε για 1980 Γάλλους πολίτες που ε, εμπίπτουν στη Τζιχάτ. Υπάρχει και μια θεά ζώνη βέβαια. Για πρώτη φορά πάντως επισήμως ο Πρωθυπουργό μας, ο Μανώλ Βάρς, αναφέρθηκε στη θεά ζώνη στην ομιλία του στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις ε, του Ιανουαρίου και αναφέρθηκε σε 3.000 περίπου Γάλλους υπηκόους. Οι μυστικές, οι μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι αυτή η αξιολόγηση, αυτή η εκτίμηση μάλλον, ε, είναι το κατώτατο όριο ενός αριθμού που όλο και αυξάνεται. 5-6 άνθρωποι είναι έτοιμοι ήδη να περάσουν στη δράση στη Γαλλία, στη βία δράση. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος κύκλος ανθρώπων. Είναι αυτοί που ε, αισθάνονται συμπάθεια, όπως φαίνεται από τα κοινωνικά δίκτυα, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όπως φαίνεται από προκλήσεις ή προκλητικές ενέργειες απέναντι στα όργανα του νόμου. Πρόκειται για σαλαφιστές Πρόκειται για ανθρώπου που έχουν υιοθετήσει έναν τρόπο ζωή που απάδει από τον συνηθισμένο τρόπο ζωή της Γαλλίας ή της Ευρώπης. Ε, είναι πολύ διαφορετικός ο δικό του τρόπο ζωή από τον δικό μας. Και επίση ε, η θέση του είναι πολύ αφήσιμη, ακόμη και απέναντι στη ριζοσπαστική βία. Δηλαδή δεν την ενθαρρύνουν κραυγαλαία και κατηγορητά, αλλά ούτε την καταδικάζουν. Αυτός είναι ο δεύτερος κύκλος ε, με δεκάδες χιλιάδες άνθρωπα που ε, αισθάνονται κάποια συμπάθεια απέναντι σε τέτοιες ισλαμιστικές ε, και ριζοσπαστικές οργανώσεις. Και αυτά τα φαινόμενα ανησυχούν πολύ τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ποιες είναι οι αιτίες αυτής της απώλειας των σημείων αναφοράς που είναι το θεμέλιο της ριζοσπαστικοποίησης. Γιατί η βάση της ε, ριζοσπαστικοποίησης, είναι η απώλεια των σημείων αναφοράς, ε, η καταβαράθρωση αυτών των σημείων αναφοράς που κρατάει εδώ και χρόνια. Το ρόλο της παιδείας είναι πολύ σημαντικός, αλλά πέραν του σχολείου έχουμε τις υπηρεσίες υγείας, ε, το ρόλο των εργοδοτών, ακόμη και των οργάνων της τάξης που προσπαθούν να γεφυρώσουν τα εκπαιδευτικά κενά, γιατί έχουμε εκπαιδευτικά κενά και στο σχολείο, γιατί όλο και περισσότεροι νέοι σήμερα δεν έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας, λεξιλόγιο, σύνταξη, ορθογραφία. Αλλά επίσης έχουμε και πολλά κενά στους κανόνες της, ε, της κοινή ζωής. Όλο και περισσότεροι νέοι έχουν προβλήματα συνέπειας, αυτοελέγχου, ευγένειας. Το θέμα είναι ότι και η δυσκολία σε πολλές ε, περιοχές, σε πολλά διαμερίσματα, οι σύλλογοι προσπαθούν να γεφυρώσουν αυτά τα κενά. Είναι ακριβώς τέτοιοι σύλλογοι που ε, ε, προωθούν αυτή την, την, το διαχωρισμό των κοινοτήτων. για παράδειγμα, δείτε τι κάνουν οι αδερφοί μουσουλμάνοι, πόσο κοινωνική δραστηριότητα έχουν. Εκεί δίνουν περισσότερη έμφαση στην συμμετοχή στην κοινότητα και όχι στην έννοια της, της γαλλικής ταυτότητας ή της ευρωπαϊκής ταυτότητας προτείνουν με βάση ε, θρησκευτικό χαρακτήρα ένα άλλο πλαίσιο που αντικαθιστά το πλαίσιο που θεσπίζει η γαλλική νομοθεσία και η κοινοτική νομοθεσία, η ενωσιακή νομοθεσία. Επίσης, ε, να αναφερθώ σε κάτι που λέμε πολύ συχνά και που δεν στέκει. Γιατί πολύ συχνά ακούω ότι η ριζοσπαστικοποίηση οφείλεται στον κοινωνικό ή στον οικονομικό υποβιβασμό, στα οικονομικά προβλήματα και τι δυσκολίε. Αυτό το επιχείρημα το χρησιμοποιούν πολύ. Αλλά είναι ανεδαφικό αυτό το ε, επιχείρημα. Γιατί στην Γαλλία το 80% των οικογενειών είναι ε, από το Μαγκρέπ, ε, αλλά ένα μεγάλο τμήμα ανήκει στην γαλλική μεσαία τάξη. Πολλά παιδιά δημοσίων υπαλλήλων προσιλητίζονται στο Ισλάμ και ριζοσπαστικοποιούνται. Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κοινωνικό υποβιβασμό, για οικονομικό υποβιβασμό. Επίσης, ένας δανός ερευνητής είπε ότι αν ο οικονομικός υποβιβασμός έχει νόημα σε κάποιες χώρες, δεν ισχύει αυτό το επιχείρημα για τη Δανία, γιατί η Δανία είναι μια ευλογία. Δεν υπάρχει ούτε δυστυχία εκεί, ούτε φτώχεια, ούτε κοινωνικός αποκλεισμό, Το σχολείο υγεία είναι ε, δωρεάν οι άνεργοι λαμβάνοντα ψηλά επιδόματα ανεργίας και όμως η Δανία μαζί με τη Γαλλία είναι από τις χώρες που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό τζιχαντιστών. Είναι αρκετά απεσιόδοξε οι προοπτικές στη Γαλλία για τη φορά της εξελίξης αυτής της πληθυσμιακής ομάδας και τη δυνατότητα να μετέλθει βίας στο μέλλον. Για παράδειγμα, ε, έχουμε σε πολλές ε, γιάφκες, ε, μεγάλο αριθμό όπλων, καραμπινών, ε, εκτοξευτών πυράβλων και ούτω καθεξής. Και αυτό ανισχύει πολύ τις αρχές, γιατί σε περίπτωση κλιμάκωσης βίας μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Η σημερινή συζήτηση, κυρία Πρόεδρε, είναι απόδειξη ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα προσπαθούν να βρουν λύσει στο φαινόμενο. Α μην ξεχνούμε όμω ότι η βάση τη στρατολόγηση των ριζοσπαστών είναι μια ρητορική που χρησιμοποιούν κάποιοι κακοπροαίρετοι και που προσπαθεί να πείσει τους νέους ότι οι δικές μας αδυναμίες και η κατάληψη των αξιών μας θα πρέπει να γίνει και να αντικατασταθεί από τις αρχές και τις αξίες του Ισλάμ. Γι' αυτό προτείνεται στους νέους μια περιπέτεια με συγκεκριμένες αξίες, με το επιχείρημα ότι εμείς πια δεν έχουμε αξίες, ούτε μπορούμε να τις υπερασπίσουμε τις αξίες μας. Οπότε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Η στρατολόγηση, ο προσιλητισμός έχει μαζικές διαστάσεις στα σχολεία, στα τζαμιά, στις φυλακές. Ένα τρίτο της ρωσιστικοποίησης στη Γαλλία γίνεται στα τζαμιά, παρόλο που δεν το λέμε φωναχτά στη Γαλλία γιατί δεν είναι πολιτικός ορθό. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Θα πρέπει να επαναφέρουμε την πυγμή και ένα πλαίσιο στεναρό. Μόνο δείχνοντας πυγμή θα ανακτήσουμε τις αξίες μας ε, για τις οποίες είμαστε περήφανοι. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και να διατρανώσουμε τις ε, ε, ιουδοχριστιανικές μας ρίζες, να εσταλάξουμε τον, το σεβασμό της εξουσίας, της ισότητας των φύλων, τη ύπαρξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια και την κουλτούρα του αποτελέσματο και όχι απλώ να περιμένουμε, στην Αθηνά και χειρακίνη. Επίση, να επιμείνουμε στην ανάγκη τη προοδευτικότητα τη εκμάθηση, ώστε οι νέοι να αποκτήσουν σταδιακά και σιγά σιγά τα εφόδια και μετά να μπορούν να περάσουν τη συζήτηση και να αναπτύξουμε και το συλλογικό πνεύμα, για παράδειγμα ρόλο του αθλητισμού. Εν κατακλείδη, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σας ε, αναφέρω δύο περιστατικά πολύ ανησυχητικά που μου διηγήθηκαν πρόσφατα τις δύο τελευταίες εβδομάδες κάποιοι γνωστοί και να σας προτείνω και κάποιες ε, δράσεις. Για παράδειγμα, ένας Γάλλος καθηγητής, καθηγητής γαλλικών, φιλόλογος, ε, που μάλιστα είναι σε ένα από τα πιο δύσκολα προάστη της Γαλλίας, που πήγε εθελοντικά εκεί, 45 ετών, πολύ ενθουσιώδης. Πριν από λίγες μέρες ένας νέος από το Μαγκρέμπ πήγε και τον βρήκε και τον ρώτησε «Πείτε μου, κύριε καθηγητά. Είναι αλήθεια ότι θα έχουμε εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία. Και ο Καθηγητή του απαντά, μα τι λέτε, ποιο το είπε. Ε, εγώ αυτό ακούω, λέει, ότι θα γίνει εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Γάλλων και Μουσουλμάνων. Οπότε ο καθηγητή ευνηδιασμένο του απαντά: Όχι, μα εγώ είμαι φιλόλογο. Εδώ στο σχολείο διδάσκουμε ότι θα πρέπει να διαβιούμε ειρηνικά, αρμονικά, να έχουμε διάλογο μεταξύ μα. Και ο νέο, κοιτώντα το προ... προκλητικά, του κόβει το λόγο και του λέει: Ναι, αλλά αν γίνει εμφύλιο πόλεμο στην, στην Αγγλία και στη Γαλλία, και ε, το πιο εύκολο θα είναι να σε σκοτώσω από τώρα. Αν μια ψυχή είναι να βία. Και μάλιστα το αυτοκίνητο του καθηγητού αυτού πυρπολήθηκε την περασμένη χρονιά. Πραγματικά ο άνθρωπο σοκαρίστηκε και ε, ένιωσε μεγάλη απεσιοδοξία μετά από το περιστατικό αυτό. Επίση, δεύτερο περιστατικό, 12 Οκτωβρίου το χωριό Σαλόν Σαμπάνι, που το γνωρίζουν μόνο οι κατοικοί του. Ένας νέος ε, μαθητής ηλικίου έφτασε λίγες μέρες μετά τη ριζοσπαστικοποίησή του με ένα πιστόλι airsoft ε, και το έστρεψε προς, ε, προς τον καθηγητή του και, και μάλιστα ε, εκπυρσοκρότησε κατά του καθηγητή και όταν το συνέλαβαν είπε στους αστυνομικούς ότι σκοπός του ήταν να σκοτώσει τον καθηγητή του και μετά τους αστυνομικούς πήγαν να το συλλάβουν γιατί ήθελε να πεθάνει ως μάρτυρας. Είναι ανησυχητικά όλα αυτά. Αλλά αυτό είναι το σχέδιο του ριζοσπαστικού Ισλάμ που έχει ρίζες πια ακόμη και στο σχολείο και στην εκπαίδευση. Και πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να σας κάνω και μερικές προτάσεις πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι κάτω χώρες, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, άρχισαν να συνειδητοποιούν την αποτυχία της ε, πλήρως πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ε, αυτό που λέμε στον Καναδά, για παράδειγμα, κάποιες λογικές προσαρμογές, κάποιες, κάποιους αμοιβαίους συμβιβασμούς ε, και η υπεροχή τη κουλτούρα των νεόφερτων, ει βάρο τη δική μα οδήγησε στη δημιουργία προβλημάτων, ρηγμάτων, στην απώλεια των σημείων αναφορά, γιατί όσοι έρχονται στη Δύση και είμαστε πρόθυμοι να του υποδεχτούμε, θα πρέπει να νιώσουν ότι έχουμε και εμεί δικέ μα αρχέ, αξίε και σημεία αναφορά. Μόνο όταν δείξουμε πυγμή στι αξίες μα θα μπορέσουμε να εντάξουμε στις κοινωνίε μα και του υπόλοιπου. Η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έγινε με καταπληκτικές βάσεις το 1950 μετά από δύο μακελιά μέσα σε 20 χρόνια που ρήμαξαν την Ευρώπη. Χρησιμοποιείται αυτή η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τους φανατικούς ως επιχείρημα για να υποσκάψουν τα ίδια τα δικαιώματα της ε, σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαίωμα της ανεξαθρησκείας, της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας συνείδησης. Ε, αυτό κάνουν στο ζούντο. Ο μικρός όμως που χρησιμοποιεί την ε, δύναμη του μεγαλόσωμου για να τον ανατρέψει. Αυτό κάνουν και αυτοί οι Ισλαμιστές. Οπότε αν εμείς και αν εσείς αν οι δικαστές, οι πολιτικοί θύνοντες δεν αντιληφθούν τη σοβαρότητα της απειλής, τότε η κοινωνία μας κινδυνεύει να καταρρεύσει. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τα προηγούμενα που μας έχει διδάξει η ιστορία. Αυτά μπορούν να συμβούν πολύ γρήγορα και η κλιμάκωση να έρθει πολύ γρήγορα σε λίγους μήνες και μερικές φορές και σε λίγες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, για τη σκληρή διαδικασία για τα σκερά που γιατί οπωσδήποτε αυτά όμως ε, έχουν ε, ρίζες πραγματικότητα και στη Γαλλία και όχι μόνο οπότε πρόκειται για κάποια πρόκληση που μας οδηγεί να σκεφτούμε ότι έχουμε κάποιες κοινέ αξίες ε, παρά την πολιτιστική πολυμορφία οπότε θα πρέπει να έχουμε τέτοια προσέγγιση ειρηνική αλλά αναπόφευκτα έτσι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα συμμεριζόμαστε τις ε, ανησυχίες σας. Ε, ακριβώς έχουμε μεγάλη πρόκληση μπροστά μας και άρα θα πρέπει να εξοπλιστούμε για να την αντιμετωπίσουμε. Και τώρα για να κλείσει τη συζήτηση θα δώσουμε τώρα τον λόγο στον κύριο Μπέργκερ από την ε, UNESCO ή Μπερζέ. Οπότε έχετε το λόγο κύριε. Κυρία Σίλβια Κώστα, Κυρία Πρόεδρε, εξότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Αυτό το ζήτημα αφορά την UNESCO και τα 195 κράτη-μέλη της. Για να δούμε τι προοπτικές έχει το ζήτημα. Είναι σαφές ότι κανείς δεν γεννιέται ριζοσπάστη της αριστεράς ή της δεξιάς. Οι άνθρωποι μεγαλώνουμε στο ιστορικό γίγνεσθε και θα πρέπει να δούμε το πώς είναι δυνατόν να ριζοσπαστικοποιηθούν και να γίνουν επιθετικοί ιδίως μέσα σε κάποια συγκυρία όπου έχουμε έλεγχο του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης από πολεμοκάμπυλους. Να για να δούμε τώρα πώς θα καταφέρουμε τις διαφάνειες. Okay, I think I have to ask uh, the people operating the computer because this doesn't work. Α, για να το κάνω από τον υπολογιστή γιατί το remote control το λέω. Για να δούμε τώρα διαδικασίες της είναι σαφές ότι δεν γεννιούνται αλλά γίνονται ε, ριζοσπάστοι άνθρωποι ε, δια της ε, πυθούς και έτσι αναλαμβάνουν ε, ένοπλη, συγγνώμη, βίαιη δράση και έτσι ταυτίζονται και οδηγούνται έτσι στην ανάληψη δράσης Επομένω αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστο από πλευρά πνευματική οικονομική, πολιτιστική για την κοινωνία. Και αυτό το οποίο κρύβεται από πίσω είναι αυτή ε, η, η ταύτιση. Οπότε ε, το επόμενο που να δούμε είναι το θέμα τη χρήση των μέσων ε, επικοινωνία και άλλων μεταβλητών. Γιατί συζητήσαμε τι γίνεται με τα σχολεία, τι γίνεται με τι οικογένειε, τι φυλακέ κλπ. Το σημαντικό επομένω είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι τα μέσα είναι μέρος ενός συνόλου. Και δεν θα πρέπει την προσέγγισή μας να την ε, εστιάζουμε μόνο στα, στα τα οποία αυτά προβάλλονται. Άρα θα πρέπει να έχουμε μια ε, σφαιρική αντίληψη των αιτίων και αποτελεσμάτων ή αντιδράσεων. Τι διακυβεύεται σε αυτή την ε, προβληματική για την UNESCO αλλά και για το δικό σας κοινοβούλιο το θέμα είναι η ελεύθερη έκφραση. Γιατί όπως γνωρίζουμε υπάρχει το δικαίωμα του να αναζητεί, να λαμβάνει και να διαδίδει κάποιος ε, πληροφορίες και ιδέες. Και έχουμε βέβαια κάποιους περιορισμούς του δικαιώματος στο άρθρο 28 αυτής της ε, διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και λέμε ότι μπορεί να υπάρξει περιορισμός αυτού του δικαιώματος στο άρθρο 20 αυτής της ε, σύμβασης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τι προβλέπετε. Ότι τα κρατημέλη Μπορούν να περιστείλουν αυτές τις ελευθερίες. Όμως το θέμα είναι ότι στην περίπτωση ριζοσπαστικοποίησης εύκολα μπαίνουν ταμπέλες και θεωρείται κάποια έκφραση ότι πρέπει να υπόκειται σε περιστολή. Και δεν είναι για εκφράσεις ριζοσπαστικές. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, πώς θα αποφύγουμε το να αντιδράσουμε δυσανάλογα και υπερβολικά σε κάποια λεκτική έκφραση ακόμα και όταν είναι προκλητική. Να μην αντιδράσουμε περιβολικά και έτσι να περιστύλουμε την ελευθερία της έκφρασης. Στην εισήγησή μου θα συζητήσω σε τέσσερις άξονες, πρώτα-πρώτα τα μέσα ενημέρωσης, να προβληματιστούμε για το τι εννοούμε και κατόπιν να πάμε στην επίπτωση και στα αποτελέσματα και κατόπιν να πάμε στο έργο που επιτελεί σχετικά η UNESCO. Και κοιτάξτε εδώ, Κάπως απλοποιημένο είναι αυτό το σχήμα, αλλά είναι καλή αφετηρία γιατί τα μέσα δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά περισσότερα. Και εδώ στη μέση έχω τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Τα βάλα στη μέση. Γιατί αυτά τα μέσα είναι ιδιαίτερα προσφυλή στην νεολαία. Που είναι πολύ ευάλωτη στη ριζοσπαστικοποίηση. Όμω υπάρχουν και άλλα ε, μέσα εκτό από τα κοινωνική δικτύωση, τα ειδησιογραφικά λέει αριστερά που δούμε στη γνώση και δεξιά τα της ε, ψυχαγωγίας που δρούν στο θυμικό, στα συναισθήματα. Για να δούμε τώρα τι δύο κατηγορίε προ τα αριστερά, κοινωνική δικτύωση και ειδησιογραφικά. Είπαμε στην επόμενη διαφάνεια, τα ειδησιογραφικά παίζουν κάποιο ρόλο, Ιδίω όταν είναι αξιόπιστα γιατί αν θεωρούνται προπαγανδιστικά δεν αποδίδουν. Τα μέσα κοινωνική δικτύωση, εάν δεν διέπονται από διαλογική δράση, επίση δεν έχουν ε, αποτέλεσμα. Πάμε τώρα εδώ να δούμε αυτό που θέλω να σας τονίσω ότι δεν πρόκειται για δύο διαφορετικούς κόσμους. Αυτό που γίνεται ε, στα μέσα, τα ειδησιογραφικά συμβαίνει στις κοινωνικές δικτύωσεις και το, τα μεν ε, επιδρούν στα δε. η γνώση επηρεάζεται πάρα πολύ από τα ειδησιογραφικά μέσα και επίσης επιδρά με τις άλλες αλλά και επηρεάζεται από το μέσα κοινωνική δικτύωσης που δημορφώνουν συμπεριφορές. Για να δούμε τώρα όλα αυτά, τι σχέση έχουν με τη συμπεριφορά του κόσμου. Υπάρχει αυτό που λέμε στα αγγλικά KAP δηλαδή γνώση, συμπεριφορά, δράση. Δηλαδή είναι ο εγκέφαλος, η καρδιά και τα χέρια κάνουν το διαχωρισμό εύκολα τι έχει σχέση με το μυαλό, τι έχει σχέση με τα χέρια, αλλά αυτό δεν είναι ευθύγραμμο, δεν είναι, ε, δεν είναι μονόδρομος, γιατί είναι δυνατόν η γνώση να διαταράξει την συμπεριφορά σε εισαγωγικά να διαταράξει και γι' αυτό και η δυσιογραφία είναι σημαντική, είναι δυνατόν να προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα δικτύωση, αλλά και αντιστρόφως. Τα μέσα δικτύωση μπορεί να οδηγήσει σε επιστράτευση αλλά και σε αντίδραση κατά αυτής. Βλέπουμε επομένω ότι υπάρχει άλλη λεξάρτηση αυτών των μεταβλητών. Όμως, όσον αφορά την κατανόηση τουλάχιστον αυτών των μεταβλητών, είναι διακριτές μεταξύ τους. Παραπέρα. Τι γίνεται με την ριζοσπαστικοποίηση και τις προσπάθειες για ανάσχεση αυτής. Εδώ έχουμε ε, διαφορετική ποιες μορφές έντασης, ε, έντονα, πιο ε, έμεσα κλπ. Γιατί το κάθε μέσο ε, συντελεί σε διαφορετικά αποτελέσματα. Τώρα έχουμε ας πούμε για τα ισχυρά αποτελέσματα, είναι βραχυπρόθεσμα τα συναισθήματα και οι λιγότερο, οι λιγότερο ισχυρές και αποτελέσματα οδηγούν σε αλλαγή της συμπεριφοράς. Για να δούμε τώρα κάτι άλλο όλα αυτά εμπλέκονται και ενεργούν από κοινού. Γιατί έχουν γίνει έρευνες και έχουν καταδείξει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα μία δεν αλλάζουν αλλά ενισχύουν κάτι. Γιατί υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που επιδρούν επί της ζωραστικοποίησης Το θέμα είναι για να ανασχέσουμε αυτή την τάση πρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Άρα το θέμα είναι περίπλοκο. Για να δούμε τώρα τα άλλα, τα έμεσα αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτού του είδους τις ροές με περισσότερες φάσεις και διαβήματα Και οι οικογένειες, οι δάσκαλοι, αυτοί που δημορφώνουν την κοινή γνώμη, διαμορφώνουν κατά πολύ την κατάσταση αυτή μέσα από τα media, μέσα από τα μέσα. Το, επίσης κάτι άλλο που διαμορφώνεται είναι το να ξέρουμε ότι ένα θέμα είναι σημαντικό. Αυτό δεν καθορίζει το πώς θα αντιδράσουμε στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά το να γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό. Οπότε πάμε τώρα στα βαθύτερα αποτελέσματα. Η κουλτούρα των μέσων ενημέρωσης, των media ομάδες, ολόκληρες κοινωνίες ζουν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον των μίντια, των μέσων. Και έτσι διαμορφώνεται η ταυτότητα, ο ρόλος, ο υποκειμενισμός. Γίνεται κάποιος εθνικιστής ή ε, γίνεται μάρτυρας ή παίρνει τον νόμο στα χέρια του ή ε, γίνεται επαναστάτης νέος ή έφηβος. Να, τι φέρνει η κουλτούρα των media. Επίσης, έχουμε κάποιο είδους πλαίσια που καθορίζουν τι είναι κλασικό και τι είναι περιθωριακό. Τι είναι καθιερωμένο και τι είναι εξαιρετική φύση. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι όλα αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να συντείνουν στην ζωσπαστικοποίηση ή όλα αυτά μπορούν να την ανασχέσουν. Δεν μπορούμε να πούμε απλά ότι είναι ένας μονόδρομος και ότι το σχήμα αυτό είναι απλό. Πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει μαϊκή συνταγή για το τι μπορεί να κάνει κανείς. Θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός ενεργειών όπως και, και αποτελεσμάτων και να καταλάβουμε ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ε, μακρόπνο, Άρα θα πρέπει κανείς να κάνει κάτι για τη ριζοβαστικοποίηση πριν ξεφύγει του ελέγχου. Για να κοιτάξτε εδώ πέρα τέσσερα στοιχεία του τι γίνεται. Το να μπλοκάρει, να αφαιρέσει, να ξεριζώσει, μετά έχουμε τον διαπολιτικό διάλογο, μετά έχουμε τα αντιπιχειρήματα και μετά έχουμε την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των μίντια. Για να δούμε. Πρώτα πρώτα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η προστασία έτσι μπλοκάρουμε ένα περιεχόμενο, ιδίω του ίντερνετ. Οπότε μειώνεται ο ερθισμός, το κίνητρο. Δεν έχουμε λάβει στη φωτιά κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, τα... αυτό το, να περιστήλουμε το ίντερνετ δεν αποδίδει πάντοτε. Πάμε παρακάτω. Όμως, κοστίζει πολύ να υπάρξουν τέτοιου είδους περιορισμό στο Ιντερνετ και για τον ιδιωτικό και για το δημόσιο τομέα. Γιατί όταν μπλοκάρουμε κάτι στο Ιντερνετ, τότε έχει κίνητρο άλλο να ψάξει το περιεχόμενο αλλού. Όριο στο περιεχόμενο σημαίνει ότι, ότι κάποια στοιχεία του Ιντερνετ πάνε στο βαθύ Ιντερνετ. Οπότε η προστασία είναι ένα μέσο αντίδραση, αλλά έχει κάποια όρια. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι που δημιουργεί η προστασία. Μπορεί κανείς να ε, εξοκύλει σε κάποιο είδους λογοκρισία. Επίσης, είναι δυνατόν κάποιοι ιδιωτικοί φορείς μπορεί να γίνουν ε, και να υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις και πριν κάνετε δημοσίευση. Το ρίσκο αυτό μπορεί να περιοριστεί γιατί θα πρέπει τα κράτη να εξισορροπήσουν τα δικαιώματα με την ε, ασφάλεια και από την άλλη μεριά χρειάζεται η διαφάνεια, η ε, ανεξαρτησία και η δυνατότητα προσφυγή στη δικαιοσύνη. Βλέπουμε επομένω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν κάποιε κρατικέ από τα Ηνωμένα Έθνη και θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη ευαισθητοποίηση. Για να δούμε παρακάτω. Και από πλευρά ε, εμπορική και από πλευρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ λέμε τι γίνεται πέρα από τις πρωτοβουλίες της προστασίας. Κανόνας θα πρέπει να είναι η ελεύθερη ροή. Να μπορεί ο κόσμος να επιλέξει και να κρίνει. Άρα θα πρέπει να τηρεί κανείς τα διεθνή πρότυπα για τον περιορισμό του δικαιώματος λόγου και να υπάρχει και κάποιο είδους ε, ετοιμότητα. Και βάζουμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι όσον αφορά την προστασία. Οπότε κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε σαν ε, μέσο προστασίας είναι η χειραφέτηση. Δηλαδή κανείς να ενημερώνει και να δημιουργήσει συνειδητοποίηση για όλα τα επίπεδα επιρροής. Θα πρέπει ο, κάθε, το κάθε άτομο να μπορεί να έχει την ταυτότητά του υπό έλεγχο και να είναι συνειδητοποιημένο κοινωνικά, να καταλάβουν τα μέσα, να ξέρουν πότε υπάρχει χειραγώγηση. Οπότε γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους να καταλαβαίνουν τι γίνεται με τα μέσα, τι ρόλο παίζουν, πώς επηρεάζουν και επομένως ε, να ξέρει κανείς τι θα πει διαπολιτιστικός διάλογος. Τρίτη πολιτική μπορούμε να έχουμε είναι ε, να προτάσουμε ενεργά κάποια αντιεπιχειρήματα. Και έτσι ο κόσμος οι να αντιστέκονται στα μηνύματα μίσους. Διάλογος και όπως λέει κάτω-κάτω η διαφάνεια να υπάρχει μια ζώνη περιοχή σεβασμού. Και να αποφεύγει κανείς όταν δεν χρειάζεται τη συναισθηματική φόρτιση. Επίσης, προσοχή για τους κινδύνους ε, αυτών των αντιεπιχειρημάτων ότι καμιά φορά για να δούμε τι λέει παρακάτω. Ότι κάποια φορά γίνεται boomerang αυτή η πολιτική. Επίσης, όταν έχουμε την ενημέρωση, ε, αρχίζουμε να υποτιμούμε, να αμαυρώνουμε τα μέσα. Και οι σχετικές εκστρατείες δεν θα πρέπει να θεωρούνται δημοσιογραφία. Γιατί θα πρέπει η δημοσιογραφία να παραμείνει αξιόπιστη και να μπορεί να έχει τη λειτουργία της ε, ε, μετάδοσης της γνώσης. Επίσης, κάτι για τα μέσα καθε αυτά. Όπως είπαμε τα ειδησιογραφικά μέσα δεν είναι σε διαφορετικό κόσμο, διαφορετικό σύμπαν σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές φορές ε, βέβαια μπορεί να έχουν τα σπέρματα κάποιας ε, αμφισβήτησης και να στρέψουν ε, ένα κομμάτι της κοινωνίας έναντι των υπολείπων ή θα πρέπει βέβαια να ε, εκθέτει κανείς τους κινδύνους της ε, βίας και χρειάζεται πλουρισμός στα μέσα είναι δυνατόν κανείς να βρει νέες αφηγήσεις και βοηθά έτσι την νεολαία. Τώρα το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι τι κάνει η UNESCO. Έχουμε ένα σωρό ε, δημοσιεύσεις κάνει στο βάθος της αίθουσας μπορεί να τα βρείτε, να ρίξετε μία ματιά και να σας τα πω αυτά γρήγορα γιατί τελειώνει ο χρόνος μου. Αλλά ξεκινήσαμε με αυτή, αυτή την ρίση της ε, διευθυντήριας κυρίας ε, Μπόκοβα ότι αυτό το οποίο είπε είναι το εξής που θα πρέπει να έχει η νεολαία τις ε, δεξιότητες, την γνώση και τις αξίες για να αντισταθεί στη ζωαστικοποίηση. Οπότε πολλές μεταβλητές εδώ μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η χειραφέτηση. Δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Οπότε έτσι κανείς μπορεί να σχέσει την ζωοπαστικοποίηση και επίσης θα πρέπει να δουλέψουμε ε, πολυκλαδικά το είπε με τα μίντια, με ε, τα πολιτιστικά, με την παιδεία, με την κοινωνική επιστήμη. Εμείς επί τόπου έχουμε ε, υπαλλήλου μας, ακριβώς και που υπάρχει το πρόβλημα. Και συνεργαζόμαστε και με άλλους διεθνείς ε, φορείς που καταβάλουν και αυτή ε, προσπάθεια. Θέλουμε επομένω έτσι να αναδείξουμε το θετικό ρόλο των νέων γυναικών αλλά και ανδρών στην αντίσταση κατά της ζωοσπαστικοποίηση. Τώρα θα σας παραλείψουμε κάποιες διαφάνειες. Πάμε στο επόμενο slide που λέει για την κατάληξη, το αποτέλεσμα της προσπαθειάς μας. Πρώτα-πρώτα, ε, για τη γνώση. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι υπερβολικά περίπλοκα και, και για τα μίδια θα πρέπει επομένως να δούμε ότι μόνο με κατανόηση μπορεί κανείς να καλύψει όλα αυτά τα ζητήματα. Επίσης ε, δυνατότητες, δραστηριότητες και οι νέοι να καταλαβαίνουν μεν το πρόβλημα αλλά επίσης να είναι στέζε. να αντιτάξουν, να αντιταχθούν σε αυτή την αρνητική επιρροή. Παρακάτω έχουμε κάποιες εκστρατείες ε, για να ενημερώσουμε τους νέους, ώστε να εμπλέξουμε εκεί τα μέσα της ενημέρωσης και να έχουμε καινούριου χώρους για να καλύψουν αυτά τα νέα μέσα, κυρίως σε συγκεκριμένες ε, ε, κοινότητες στην κοινωνία. Με λίγα λόγια. Αυτά κάνει η UNESCO, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μας απασχολεί, οπότε να δηλώσω την παρουσίασή μου. Για να δούμε. Έγινε διάγνωση των αποτελεσμάτων των, των αλλά επίσης είδαμε και πώς ε, κανείς μπορεί να αντιδράσει. Είδαμε επίσης πώς είναι αυτή η σφαιρική ολοκληρωμένη ε, αντίδραση της ε, UNESCO στο πρόβλημα της ριζοσπαστικοποίησης. Οπότε, το τι θα κάνουμε. Νομίζω, στον τελευταία αυτή διαφάνεια, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τον ρόλο των μίντια στην ριζοσπαστικοποίηση. Οι πέντζα σκοπάζεται υπάρχει. Και είπαμε, πάμε τι γίνεται με την επιρροή των ε, μεταναστών. Γιατί θα πρέπει να προβλέψουμε το μέλλον. Γιατί θα έχουμε κομμάτι της κοινωνία που θα είναι κατά των μεταναστών και θα υπάρξουν και κάποιες εκφράσεις αυτής της τάσης. Είπαμε ότι χρειάζεται σφαιρική προσέγγιση αλλά με ό,τι κάνουμε να μην υπονομεύσουμε τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρωπότητας. Πολύ σημαντικό αυτό για την κοινωνία σας για την, σύνομαι, για την Επιτροπή σας όσον αφορά τα οπτικοακουστικά και τα πολιτιστικά. Επίση, χρειάζεται φυσικά υποστήριξη οικονομικών πόρων για αυτές τις προσπάθειες. 40 εκατομμύρια το μήνα κερδίζει πουλώντας πετρέλαιο το Ισλαμικό κράτος. Αλλά έχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης. 40 εκατομμύρια δεν είναι δυνατόν να μην πρικοδοτήσουμε αρκετά την πρωτοβουλία κατά της ζωσβαστικοποίησης. Όσο καθυστερούμε τόσο μεγαλώνει το πρόβλημα. Και θα γίνεται όλο ένα και πιο ακριβό το να πρικοδοτήσουμε την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ε, ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ όλους σας. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Και βεβαίως οι εμπειρογνώμονες μας θα απαντήσουν στη συνέχεια. Παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί έχει προχωρήσει η ώρα. Παρακαλώ. Ε, κυρία Βόρτ. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να μιλήσω, ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι Εκπονώ εγώ μια πολύ σημαντική έκθεση ε, για την Επιτροπή μας, για το διαπολιτισμικό διάλογο, την ε, ε, πολυμορφία, την κοινωνία και το έχουμε συζητήσει με τους σκιώδεις συγητές. Όλα αυτά τα θέματα που αναφέρετε και εσείς τα βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας. Όχι μόνο στην Επιτροπή Πολιτισμού και σε άλλες επιτροπές. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι εκτίμησα πάρα πολύ τα όσα μας είπατε Σάρα προηγουμένως ε, είσαι συμπατριώτησά μου και κάνεις καταπληκτική δουλειά. Προηγουμένως ε, είχα πάει σε μια συνέντευξη στο Πρασίνο να ε, μιλήσω. Ε, χαίρομαι που εδώ ε, είσαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ εκπροσωπώ τη Βορειοδυτική Αγγλία. και προέρχομαι από ένα δημιουργικό παρελθόν, ας πούμε, καλλιτέχνης όλη μου τη ζωή. Συνεργάζομαι με ανθρώπους των κοινοτήτων αυτών και για μένα αυτό το θέμα δεν είναι ε, η πολιτική μου δραστηριότητα. Όλη μου τη ζωή με θέμα τα ασχολούμαι, η δουλειά μου. Και ε, ε, ο πολιτισμός δεν είναι κάτι το δεδομένο, δεν είναι κάτι το καθυλωμένο. Δεν ισχύει αυτό, ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει, ούτε στο μέλλον ο πολιτισμός είναι πολλά. Εμείς έχουμε πολλαπλές ταυτότητες, δεν έχουμε μία. Και ο πολιτισμός είναι ένα τμήμα και η κουλτούρα. Είναι κάτι το οποίο ρέει συνεχώς. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τη δική σας παρουσίαση, κύριε ε, ε, Μπέργκερ, να μιλάτε για την ριζοσπαστικοποίηση με πολλούς τρόπους. Δύο εβδομάδες το καλοκαίρι ήμουν εθελόντρια στη Βοσνία και δύο από τους εθελοντές εδώ που συνεργαζόμαστε είναι παρόντες ε, για ένα πρόγραμμα Ευρωπαίων πολιτών και πήραν και το βραβείο του Ευρωπαίου πολίτη χτες. Σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν στη Στρεμπρενίτσα συζητήσαμε ε, αυτό που έκανε ο Άντρες Μπρέβικ στην Νορβηγία. Και ποια είναι η ριζοσπαστικοποίηση της δεξιάς. Δεν το συζητάμε ποτέ της πολιτικής δεξιάς. Συνεχώ μιλάμε για τη ριζοσπαστικοποίηση, λες και είναι κάτι που αφορά μόνο τους μουσουλμάνους. Και θα πρέπει να θυμηθούμε και αυτά τα φαινόμενα. Ε, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο εγώ διαδήλωσα κατά του 50 του γερμανικού κινήματος και είναι και για μας μεγάλο πρόβλημα και δεν έχει να κάνει μόνο ε, με ένα ε, εθνοτικό background. Συγγνώμη που πηγαίνω, έρχομαι, γιατί πηγαίνω και σε άλλες επιτροπές και ψηφίζω και έχουμε παράλληλες συνεδριάσεις. Χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα και αυτά που είπατε θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα συγγνώμη, για τη δική μου έκθεση και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Μομπριάλ. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του γιατί μας παρουσίασε τη Γαλλία στο χείλο εμφυλίου πολέμου. Δεν ξέρω. διάβασα εγώ μια συνέντευξη του Αλέν Βίλφιν που με τίτλο «Η Γαλλία διαλύεται». Φαίνεται και στο γαλλικό τύπο να υπάρχουν τέτοιες ε, ανησυχίες. Εσείς είπατε ότι αυτή η κατάσταση οφείλεται στις αδυναμίες ε, της, ε, του γαλλικού κράτους και της γαλλικής κουλτούρας. Ποια είναι τα αίτια όμως αυτής της αδυναμίας και αυτής της κατάστασης. Ποιες είναι οι αιτίες που δεν προβάλλονται δεόντως οι αξίες μας. Επίσης, Ο κύριος Μπέργκερ μας ε, μίλησε για, για τις επικρίσεις του Μοφρέη σημαντικού στοχαστή Γάλλου του Μισελ Οφχέ, συγγνώμη και αμέσως χαρακτηρίστηκε ε, εξτρεμιστής. Μα υπάρχει πρόβλημα με την αδυναμία της κουλτούρας μας, του πολιτισμού μας να προασπίσει τις αξίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονές μας για τις παρουσιάσεις τους όσο και για τις συστάσεις τους. Νομίζω ότι στα όσα μας είπε ο κύριος από την UNESCO αναφέρθηκε στο ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω και το ρόλο των δημοσίων κρατικών μέσων ενημέρωσης. Διότι πιστεύω ότι ε, τα δημόσια ΜΜΕ είναι υποχρεωμένα να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της βίας. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε ε, να πούμε ότι είναι μια δικαιολογημένη ε, ε, μάχη και ένας αγώνας που δίνει. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Χάν, διότι οι μαρτυρίες αυτές που μας ανέφερε για τις μουσουλμάνες είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Ότι οι μουσουλμάνες είναι ίδιες κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Ότι έχουν δράσεις και δραστηριότητες κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Ε, αυτά είναι προφορίες που θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμες και θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου. Ε, σε... Και επίσης, ε, αυτό για μένα είναι φως στην άκρη του τούνελ και ελπίδα. Ελπίζω Ελπίζω να ε, σε αυτή με επιτυχία αυτή η προσπάθειά μας. Ευχαριστώ. Βεβαίω θέλουμε να μάθουμε και τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δώσουμε το λόγο. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλετε να μιλήσει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο τέλος. Θέλετε τώρα να σχολιάσουμε αυτά που ακούσαμε. Μάλιστα εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση ε, Εσωτερικών για τη διαχείριση των κρίσεων και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ε, τόσο ενδιαφέρουσα ακρόαση. Πρώτον, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δεν υπάρχει ένας και μόνο ε, τρόπος και μορφή ριζοσπαστικοποίησης. Είναι πολλές οι απειλές. Αυτό το λέει και η Ευρωπόλ στην ετήσια έκθεση που κάνει για την εκτίμηση της απειλής ε, ε, έχουμε επιθέσεις ε, θρησκευτικού χαρακτήρα στην τέταρτη θέση. Οι αποσχιστικές ομάδες και επαναστατικές έρχονται πρώτες σε επιθέσεις ή απόπειρες, δεξιά και αριστερά. Αναρχική είναι η δεύτερη και αριστερα αναρχικη ειναι δευτερη και τριτη Και ο θρησκευτικός ριζοσπαστισμός και η τρομοκρατία είναι Τέταρτος και μετά πέμπτος είναι τα μονοθεματικά όπως ανθρώπινα δικαιώματα, κατά των αμβλώσεων κτλ. Αυτά είναι τα ποσοτικά στοιχεία. Βεβαίως ποιοτικά ορισμένες ομάδες ε, τζιχατιστών, ιδιαίτερα όσοι επιστρέφουν και έχουν εμπειρία μάχης, ε, είναι πάρα πολύ κρίσιμη απειλή. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολλές πτυχές Δεύτερον, δεν υπάρχει ένα προφίλ και μοναδικό, το ακούσαμε και προηγουμένως. Δεν υπάρχει ένας χαρακτήρας. Αλλά οι περισσότεροι νέοι, που δεν είναι και τόσο νέοι κατά τα άλλα, που μπαίνουν στο τζιχάντ, έχουν πάρα πολύ επιφανειακή, επιπόλαια ε, και λεπτή θρησκευτική προέλευση. Δηλαδή, αν δούμε κάτω από την επιφάνεια, δεν είναι θέμα θρησκευτικών πεπιθήσεων, είναι αυτό που είπε η κυρία Καν. Είναι, θέλουν να δώσουν ένα νόημα στη ζωή τους. Ε, κάποια υπαρξιακά ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν. Τα είπε και ο κύριος Δεμομπριάλ. Και επίσης ε, υπάρχουν αυτοί οι ριζοσπαστές κήρυκες, ιεροκήρυκες, με απαντήσεις έτοιμες για οτιδήποτε ερώτημα έχει κανείς κοινωνικό, φιλοσοφικό, υπαρξιακό, ένταξη στην κοινωνία κλπ. Επιβεβαιώνω το αριθμητικό στοιχείο 20% των ξένων μαχητών είναι ε, προσιλητισμένοι. Δεν ήταν μουσουλμάνοι, αλλά ξοπίστησαν. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ του Ισλάμ ως πίστη, ως θρησκεία και τον Ισλαμισμό και το ριζικό Ισλάμ, το ακραίο, που είναι πρόφαση. Τηλεγραφικά τα λέγω. Ποιε είναι οι απαντήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι ε, η αλυσίδα ασφαλείας, δηλαδή ε, υπηρεσίε πληροφοριών, επιβολή του νόμου, ε, δικαιοσύνη και σοφρονιστικό σύστημα έχουν ρόλο να παίξουν πρωταγωνιστικό. Δεν είναι μόνο θέμα ασφαλείας. Η ριζοσπαστικοποίηση αφορά την ίδια μας την κοινωνία και όχι μόνο τις εγκληματικέ συμπεριφορές. Υπάρχει και ε, ε, η λεγόμενη μαλακή πλευρά της δημοκρατίας που είναι η πιο σκληρή διότι χρειάζονται μέρες, μήνες, εβδομάδες για να ριζοσπαστικοποιηθείς, αλλά χρειάζεται μισή γενιά περίπου ή μια γενιά για να γίνεις ένας φιλήσυχος φιλελληνικός πολίτης και συνειδητοποιημένος. Εμείς τι κάναμε, συστήσαμε αυτό το ε, δίκτυο με 2.000 οργανώσεις στην Ευρώπη, ε, σαν αυτή που περιέγραψε η κυρία Χάν, που εργάζονται ακριβώς στη βάση ε, στην κοινωνία για να εντοπίσουν τα αρχικά συμπτώματα. Λέγεται ένα κέντρο συνειδητοποίηση και επαγρύπνηση για τη ριζοσπαστικοποίηση. Δεν θέλω εκεί να επιμείνω, αλλά έχουν εντοπίσει καλές πρακτικές για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των πρώιμων σημείων ριζοσπαστικοποίηση. Ε, σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Βεβαίως πιστεύουμε ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι αδιαπραγμάτευτη και απόλυτη. Αλλά Υπάρχει περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο ίντερνετ και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης που, υπάρχει online έτσι και δεν θα το δεχόμασταν σε καμία περίπτωση ε, στον πραγματικό κόσμο, εδώ στο περίπτερο κάτω να τα πουλάνε. Οπότε Ποια είναι η πρόκληση να αντιμετωπίσουμε, να εντοπίσουμε μάλλον αυτή την προπαγάνδα, αυτά τα ακραία και να τα αφαιρέσουμε. Βεβαίω μετά θα φυτρώσουν άλλε ιστοσελίδε όπου ε, κόβει ένα ιστότοπο. Να αντιμετωπίσουμε ε, το περιεχόμενο, να το αφαιρούμε, όχι εμεί, οι εταιρείε οι Δεν ε, θέλουμε να επιβάλλουμε τίποτα σε κανέναν, αλλά προειδοποιούμε ε, τα social media ε, ότι ορισμένοι χρήστες παραβιάζουν τον νόμο. Και το τρίτο είναι να δημιουργούμε επαφές και πολλές. Και έχει σημασία εδώ και η ποσότητα. Ο λόγος είναι ένα προς εκατό. Δηλαδή μια μετριοπαθής φωνή αντιστοιχεί σε 100 ε, φωνές ε, προπαγανδιστικές και κηρύγματα μίσους. Και επίσης ε, το θέμα είναι να προστατεύουμε τα συστήματά μας. Και εδώ μιλώ για την ασφάλεια στον κυβερνό χώρο. Κοιτάξτε τις επιθέσεις που έχουν δεχτεί θεσμοί, όργανα, επιχειρήσεις καθημερινά, τηλεοράσεις, κανάλια κλπ και όλο και περισσότερο το θέμα είναι η πρόσβαση στο περιεχόμενο για λόγους ε, υπηρεσιών πληροφοριών και επιβολής του νόμου. Υπάρχει το θέμα της κρυπτογράφησης που είναι πολύ δύσκολο. Αν μου δώσετε ένα λεπτό, έχω ε, τη συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και εργάζονται πάρα πολύ σε αυτά τα προγράμματα ε, ανάντι και θα ήθελε και εκείνη να σας μιλήσει θα ήθελα να σας πω, συγγνώμη, ε, αλλά δεν θέλω να σας επιβάλλω ένα λεπτό. Όχι, μιλήστε όσο θέλετε. Έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε, αν θέλετε μιλήστε. Ένα λεπτό, ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα και εγώ να προσθέσω σε αυτά που είπε ο αδελφός μου μόλις ε, κάποια πράγματα από τη δική μας μονάδα που είναι αρμόδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και όλες οι παρεμβάσεις σήμερα το απόγευμα. Θα ήθελα λίγο να θυμίσω ότι οι Υπουργοί Παιδείας στο Παρίσι κατέληξαν το Μάρτιο σε μία διακήρυξη, το Μάρτιο του 2015, και είναι πολύ σημαντικό να επιστήσουμε και την προσοχή. Είναι πολύ ευρύ το πεδίο που καλύπτει βεβαίως και κυρίως ε, έχει να κάνει με τον προληπτικό ρόλο ε, της παιδείας και η προώθηση των ε, θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η διακήρυξη του Μαρτίου. Αλλά εκτός αυτού ε, πρόκειται για την ανοχή, για τη μη διακρίσεις, ε, την πολυμορφία και την άρση των αποκλεισμών. Είναι μια ευρεία λοιπόν απάντηση αυτή στην πρόληψη και να δούμε και πού συμβαίνουν όλα αυτά. Κάθε εδαφικό επίπεδο, η κάθε διοίκηση, τοπική, περιφερειακή, εθνική, ευρωπαϊκή έχει το δικό της ρόλο να διαδραματίσει. Και ε, είναι διαβίου μάθηση, δεν είναι μόνο το σχολείο και η διδακτέα ή το πρόγραμμα σπουδών. Βεβαίω το σχολείο έχει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά έχουμε την επαγγελματική κατάρτιση, έχουμε την διτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε την εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι διάφορα επίπεδα αυτά που πρέπει να μας απασχολήσουν. Πολύ σύντομα λοιπόν, τι κάνει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει συνέχεια στη διακήρυξη των ε, Παρισίων, ε, των Υπουργών Παιδείας. Δύο είναι τα βασικά που κάνουμε. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τα εφιστάμενα μέσα για την συνεργασία στην παιδεία. Από τη μια έχουμε συνεργασία σε παιδεία πολιτικής, μια ήπια συνεργασία. Ξέρετε ότι είναι εθνική αρμοδιότητα η παιδεία, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά εκεί που υπάρχει χώρος και έδαφος. Και εσύ έχουμε δύο εκθέσεις πρόσφατες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, μία και το άλλο για τις πολιτικές για την νεολαία. Αν διαβάσετε τις εκθέσεις που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο, θα διαπιστώσετε ότι ε, είναι ενισχυμένος ο ρόλος ε, της πολυμορφίας, το, ε, της συμπερίληψης και κατά του αποκλεισμού και της πρόληψης. Οι εκθέσεις αυτές μας βοηθούν λοιπόν να ασχοληθούμε ε, με βέλτιστες πρακτικές, ομάδες εργασίας, να αλληλοδιδασκόμεθα. Έχουμε θέσει ένα πλαίσιο για τη συνεργασία των κρατών μελών. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και εσείς αναφερθήκατε στις ανταλλαγές των πρακτικών. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι τα προγράμματα που έχουμε, ιδιαίτερα το Erasmus ε, Plus, που προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε ήδη από του χρόνου, το έχουμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη, πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε ήδη από τώρα διάφορες δράσεις. Κάθε είδους. Έχουμε ήδη πάρα πολύ υλικό και μπορούμε να το διαδώσουμε να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία περισσότερο μεταξύ των διαφόρων δικτύων σε τοπικό επίπεδο, ΜΚΟ και ε, κοινωνία των πολιτών. Ε, και περισσότερες ανταλλαγές μεταξύ δασκάλων, για παράδειγμα, ε, και εικονικές αλλά και πραγματικές ανταλλαγές με εκπαίδευση και ηλεκτρονική εκπαίδευση. Και επίσης προσπαθούμε να ενισχύσουμε το διάλογό μας με την ευρωπαϊκό όμω επίπεδο, γιατί διαπιστώνουμε ότι γίνονται πάρα πολλά καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά λείπει ο σύνδεσμος με τα ε, κράτη-μέλη και τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Εκεί αξίζει να υπάρχει ένα ξεχωριστό διάλογο και θέλουμε εμεί να τον ενισχύσουμε. Ξέρετε ότι έχουμε το ετήσιο φόρουμ την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη για την παιδεία και είναι προσκεκλημένα όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, Πολιτισμού στο φόρουμ αυτό. Ακριβώς για να μπορέσουμε να συναντήσουμε την κοινωνία των πολιτών έχουμε αφιερώσει και συζήτηση πάνελ για την περίοδο μετά ε, τη Συμφωνία των Παρισίων και με μεγάλη χαρά θα σας προσκαλούμε να έρθετε Δευτέρα και Τρίτη εδώ στις Βρυξέλλες σε αυτό το φόρουμ. Σας ευχαριστώ που μου αφήσετε να μιλήσω παραπάνω από ένα λεπτό. Και εμείς σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα... Α, έχουμε και άλλο συνάδελφο, ο κύριος Λιούερ ήρθε αργότερα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, προσπαθώ να συντονίσω ε, δύο επιτροπές, αυτό λειτουργεί τις περισσότερες μέρες του χρόνου και δύο-τρεις μέρες όχι, σε αυτές πέσαμε. Ε, ξέρετε ότι η ομάδα των συντηρητικών έχει πρόεδρο μουσουλμάνο που είναι φίλος και δικός μου και του καθηγητή ε, Κρασνοντέσκη και πολύ σοβαρά παίρνουμε αυτά τα πράγματα υπόψη. Μπορεί να σας εξέπληξε αυτό αλλά Μια δημοσκόπηση στη Βρετανία έδειξε ότι 27% ε, έχουν συμπάθεια με τους ε, τρομοκράτες και ένας στους 10 είπε ότι τάξιζαν οι σχιζογράφοι αυτά που έπαθαν. Ε, αυτό είναι σε μια έρευνα δημοσκόπηση που έκανε η εφημερίδα Telegraph. Οι κοινότητες αυτές λοιπόν φέρουν και εκείνες την ευθύνη τους και θα πρέπει να την επομισθούν. Εγώ αναγνωρίζω το έργο της κυρίας Καν, την οποία ξέρω και εκτιμώ το έργο της και τη θαυμάζω, αλλά πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα δρόμο που θα μας οδηγήσει στη λύση, ε, η ίδια δηλαδή η μουσουλμανική κοινότητα να αντιμετωπίσει το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης των μελών της. Σας ευχαριστώ πολύ. Βέβαια το έγκλημα δεν μπορεί να είναι λύση για έναν πολιτισμένο άνθρωπο. Είναι δικαιολόγητο σε κάθε περίπτωση. Ο κύριος Δεμομπρεάλ. Ευχαριστώ. Δεν θα απαντήσω ενδελεχώς στις ερωτήσεις σας κύριε Κρασοντέμσκι για να μην μακρηγορήσω. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι όντως η Γαλλία βρίσκεται σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Και ο λόγος είναι ότι για οικονομικούς λόγους είχαμε μαζική οικονομική μετανάστευση στη δεκαετία του 70 για να στηρίξουμε την οικονομική μας ανάπτυξη και θεωρήσαμε ότι θα εντάσσονταν ε, κοινωνικά αυτό ο πληθυσμό όπως είχε γίνει το με το προηγούμενο κύμα μεταναστών από τον Νότο και από ανατολικές χώρες. Θεωρήσαμε ότι η μαζική μετανάστευση ε, πληθυσμών δεν θα προσέκουε σε προβλήματα κοινωνικής ένταξης, γιατί είχαμε θετική εμπειρία από το παρελθόν. Βέβαια, αυτή τη φορά είχαμε διαφορετική κατάσταση, γιατί δεν ε, υποδεχθήκαμε τους ε, νέους μετανάστες με τους δικούς μας όρους και στη δική μας κουλτούρα. Και έτσι είχαμε δαιμονοποίηση και κάποιων ε, διανοουμένων που κατηγορήθηκαν ότι παίζουν το παιχνίδι του εθνικού μετόπου. Και το πρόβλημα είναι η παρέτηση ουσιαστικά των ε, γαλλικών ελίτ από το θέμα αυτό. Έτσι αφήσαμε το θέμα της μετανάστευσης, της ταυτότητας και το συναφές θέμα της ασφάλειας, το αφήσαμε να το μονοπολίσει ένα και μόνο κόμμα. Ουσιαστικά ε, απαγορεύεται, είναι ταμπού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλιώς κατηγορούμαστε ότι παίζουμε το παιχνίδι του εθνικού μετώπου της Μαρή Λαπέν. Αυτό είναι το στίγμα η ρετσινιά που κολλάμε σε όσους ε, ξεφεύγουν λίγο από το πολιτικό mainstream εδώ και ένα χρόνο. Και οπότε αφήνουμε το ακροδεξιό κόμμα να μονοπολεί τη συζήτηση και να καπηλεύεται αυτό το θέμα της ασφάλειας. Το θέμα είναι όλοι οι πολίτες, από όποια πολιτική παράταξη και προέρχονται, γιατί υπάρχουν πολίτες της ε, αριστεράς που εφορούνται από ρεπουμπλικανικές αξίες στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού που θα μπορούσαν να επαναφέρουν αυτό το θέμα. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλάει για την εφαρμογή τεχνικών μέτρων. Είναι και αυτά απαραίτητα, αλλά αλλού είναι η βάση. Θα πρέπει, βάση των μέτρων αυτών είναι η επανάκτηση των αξιών και των αρχών μας. Έτσι μόνο θα αποδυναμώσουμε τους ε, ψηφοθερικούς εξτρεμισμούς. Γιατί πού στηρίζεται η ψηφοθερία των ε, εξτρεμιστών στο ότι θεωρούν ότι θέλουν να πείσουν τον κόσμο ότι οι ανησυχίες του δεν λαμβάνονται υπόψη από τις πολιτικές ελίτ. Θα πρέπει και οι πολιτικές ελίτ να επανέλθουν σε ένα πεφωτισμένο λόγο. Έτσι θα αποδυναμώσουν τους εξτρεμιστές. Αλλά φυσικά θα χρειαστεί ίσως μισή και έως και μία γενιά για να επανέλθουμε σε μία κατάσταση πιο υγιή όπως θα έπρεπε να είναι. Τότε θα οδηγήσουμε πραγματικά σε καταβαράρθρωση του ψηφοθυρικού εξτρεμισμού. Thank you. Um, like to... Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω αυτά που ακούσα. Σε ένα πρόσφατο άρθρο εφημερίδας, ένα συνάδελφος τη κυρίας Καν ε, λέει ότι είναι σημαντικό να διδάσκονται οι μαθητές ε, και να θαρρύνονται για κριτική σκέψη και να αμφισβητούν ε, αυτά που ακούν, να ασκούν την κριτική του σκέψη για να μην τους υπαγορεύονται άνωθεν κάποιες αρχές ή αξίες. Οπότε αυτό που θα πρότεινα εγώ και θα σύστηνα στους υπουργού παιδείας είναι αυτό για να λειτουργήσει την πράξη. Η διδασκαλία της ιστορίας να αποτελέσει το αντικείμενο συνεχούς διαλόγου μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος. Στην πατρίδα μου, για παράδειγμα, όταν διδάσκουμε τις σταυροφορίες, ξεκινάμε με ένα πρόσφατο άρθρο όπου ακούμε κάποιες ριζοσπαστικές ιδέες για τις σταυροφορίες και κάνουμε το μάθημα διαδραστικά σε μια συνεχή αμφίδρομη κίνηση παρελθόντος παρόντος. Έτσι διευρύνουμε και τη συζήτηση και ενισχύουμε, ενθαρρύνουμε το διάλογο. Επίσης είχαμε την 10η Σεπτεμβρίου και τα γεγονότα. Εκεί είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε ένα ευρύ φάσμα ιστορικών πηγών και σύγχρονων και επίκαιρων και να τις αναλύουμε, να τις συζητούμε. Έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε ένα δημοκρατικό διάλογο και στις αίθουσες διδασκαλίας. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας παραγωγικός τρόπος για να συμπεριλάβουμε και τις μειονότητες στο διάλογο και να τους δώσουμε το λόγο, να τους δώσουμε φωνή και να έχουμε και μια τεκμηριωμένη συζήτηση στις αίθουσες διδασκαλίας για το τι συμβαίνει. Αυτή είναι η πρότασή μου. Uh, thank Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας πολύ ενδιαφέρουσες. Αυτό που εγώ κρατώ είναι το εξής. Η συνολική προσέγγιση, η καθολική, είναι το μόνο που μπορεί κανείς να υιοθετήσει. Υπάρχουν στοιχεία ασφαλείας, υπάρχουν στοιχεία εκπαίδευσης, υπάρχουν στοιχεία κουλτούρας και νοοτροπίας και κάθε είδους μίντια ενέχονται εκεί. Το θέμα της γνώσης και της κατανόησης που δείχνει πόσο σημαντικές είναι κοινωνικές επιστήμες. Αυτό που μας είπε η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών για τον κατάλογο των διαφόρων επιθέσεων ε, και ποια κίνητρα είχαν. Τέτοιου είδους πληροφόρηση ε, πρέπει κάποιος να σκάψει για να τη βρει, να κάνει έρευνα. Δεν ε, μα έρχεται ουρανοκατέβατη. Και η Επιτροπή Πολιτισμού στην καθολική αυτή προσέγγιση έχει να διαδραματίσει οπωσδήποτε ρόλο. Τελειώνω λέγοντας Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε όλη αυτή τη συζήτηση να θεωρείται η νεολαία απειλή αντί για πλούτος. Προσοχή. Γιατί αν δεν φέρουμε τη νεολαία στο κέντρο πολλών δραστηριοτήτων υπάρχει κίνδυνος να τη χάσουμε. Θα πρέπει να χειραφετηθούν οι νέοι για να αναλάβουν ηγετική δράση στην καταπολέμηση της ζωσπαστικοποίησης που μπορεί να προέρχεται από διάφορες κατευθύνσεις. Και σας είπα ότι φοβούμε ε, ότι υπάρχει κάτι το οποίο αναδύεται αυτή τη στιγμή. Ε, κυρία Χάν, θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με όλα αυτά που είπατε για τι διάφορε μορφέ ρίζοσπαστικοποίηση, ότι δεν υπάρχει ένα και μοναδικό προφίλ δράση. Όλα αυτά πολύ ωραία τεκμηριώνονται ε, πώς συνεργαζόμαστε με, κοινωνία των πολιτών, με την κοινωνία των πολιτών και μουσουλμάνους. Κοιτάξτε, δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε ως δίπολα όλα αυτά ε, και να πολλώνουμε τη συζήτηση. Είναι τεράστια διαφορά μεταξύ Ισλάμ και Ισλαμικού εξτρεμισμού. Οι μουσουλμάνοι δεν είναι κάτι το ομοιογενές, δεν είναι μια ομάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 3,9 εκατομμύρια οι μουσουλμάνοι που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και έχουν τεράστια πολυμορφία στην κουλτούρα, στην οτροπία, στη γλώσσα, στην παιδεία. Έχει γίνει μεγάλη έρευνα από ε, τις τοπικές αρχές και είναι λάθος να προσπαθούμε να ομοιογενοποιούμε τους μουσουλμάνους. Έχουμε και δεξιούς και αριστερούς μουσουλμάνους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ποικιλομορφία. Αν προσπαθούμε να απολώσουμε τη συζήτηση και να λέμε ότι εμείς είμαστε κάτι και οι μουσουλμάνοι είναι ο άλλος, ε, εκεί δεν πρόκειται να λυθεί η συζήτηση. Γιατί έτσι αποξενώνετε και τους ίδιους τους μουσουλμάνους που θέλετε να τους βοηθήσετε να καταπολεμήσουμε ε, την αφήγηση των εξτρεμιστών. Και εγώ μουσουλμάνα είμαι και ξέρω ότι είμαι σε διασταυρούμενα πυρά. Ε, δέχομαι απειλές από σαλαφιστές, από Ισλαμιστές κάθε μέρα, ακριβώς για τη δουλειά που κάνουμε. Ακριβώς γιατί εμείς είμαστε υπέρ των αρχών και των αξιών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έγινε μεγάλος λόγος για τις ιουδεοχριστιανικές ε, αρχές. Εγώ ούτε Εβραία είμαι, ούτε χριστιανή, είμαι μουσουλμάνα και πιστεύω στις ίδιες αρχές και αξίες δεν είναι σύγκρουση των πολιτισμών. Αυτό είναι παραπλανητικό ως υπόδειγμα. Γιατί μας το έχει διδάξει η ίδια ιστορία, ότι είμαστε Ευρωπαίοι και ευρωπαϊκές και μουσουλμανικές αξίες που υποτίθεται ότι ήταν διακριτές. Ε, είναι λάθος αυτό παράδειγμα και ψευτοδήλημα από τη μια ε, Ιουδεοχριστιανικές και από την άλλη μουσουλμανικές αξίες. Από τη στιγμή που αναδύθηκε το Ισλάμ υπάρχει αλληλεπίδραση και ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βρετανία έδειξαν οι έρευνες ότι είχαν κρίσιμη ε, συμμετοχή οι μουσουλμάνοι με τις δομές που είχαν για την απόδοση του δικαίου στη διαμόρφωση του ε, αγγλικού συστήματος. και οι μουσουλμάνοι, οι Άραβες έφεραν τον Αριστοτέλη στην Ευρώπη. Και στον 9ο αιώνα υπήρχε πολύ μεγάλη ε, διάδοση των ιδεών της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας για τις ε, μετάφρασεις στα αραβικά. Δεν είναι καθυλωμένες αυτές οι ιδέες ε, και ιστορικά δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Και επειδή ζούμε σε ένα παγκοσμιακό κόσμο, ιδιαίτερα σήμερα, όπως είπε και συνάδελφος από το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρία Γόρτ, παραμένουν ακέραιες αυτές οι αξίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε με ομάδες κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι η δική μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να συμφιλιώσουν την πίστη τους με την εθνική ταυτότητα. Και αν δεν συνεργαστούμε με ανθρώπους σαν εμένα, αν θέλουμε να τους αποξενώσουμε ή να πούμε ότι εσύ είσαι κάτι άλλο, είσαι ο απέναντι, δεν λύνεται το πρόβλημα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε, οι ομάδες ε, σαλαφιστές έχουν πολλά λεφτά. Τους χρηματοδοτούν οργανώσεις και χώρες ακόμα της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα ε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τέτοιου είδου κράτη, ενώ εμείς δεν έχουμε καλή χρηματοδότηση, ακριβώς γιατί διαδίδουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλουμε να απελευθερώσουμε τον κόσμο να χειραφετηθεί και υπάρχουν πολλοί νέοι μουσουλμάνοι που θέλουν να ακούσουν τα δικά μας μηνύματα, να τους δώσουμε τη δύναμη να το κάνουν, διψάνε να αγωνιστούν σε αυτή τη μάχη. Ευχαριστώ. Ε, Ο Πρόεδρος. Ε, μερικές λίγες παρατηρήσεις πολύ σημαντικές για να κλείσουμε. Η τελευταία παρέμβαση της κυρίας Χάνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Πράγματι, είναι εκ των όνων Να ε, μην κάνουμε ε, χονδροειδείς εκτιμήσεις για τα θέματα αυτά. η πολυμορφία είναι πολύ σημαντική όπως και στο χριστιανισμό έχουμε πολύ διαφορετικές εκφάνσεις, το ίδιο ισχύει και στο Ισλάμ. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο εσωτερικό του. Και οι αξίες εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις σε αυτόν τον κόσμο λαμβάνονται βεβιασμένα, γιατί τρέχουμε. Ο κόσμος μας αυτό είναι σήμερα. Τρέχουμε να παίρνουμε αποφάσεις και να ζούμε με ξέφρενους ρυθμούς. Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλη αυτή τη συζήτηση, βεβαίως και όλους τους συναδέλφους. Ε, ε, ρίξαμε φως σε ένα θέμα που είναι περίπλοκο, που είναι δύσκολο και επίκαιρο και σίγουρα θα απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας για πολύ καιρό ακόμα στην Ευρώπη. Θυμάστε την ε, ε, Μαλαλάου Σαχσάη που είπε ότι ένας καθηγητής, ένας μαθητής, ένα βιβλίο, ένα μολύβι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο όταν βραβεύτηκε με το βραβείο Ζαχάρα αυτά είπε αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προωθήσουμε την κουλτούρα της Ευρώπης, της επικοινωμορφίας, έτσι ώστε τα παιδιά μας θα ζήσουν σε έναν κόσμο ε, πολυπολιτισμικό. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση αυτή και η επόμενη συνεδρίαση 12 Νοεμβρίου 9 με 12.30 και 3 με 6.30 το απόγευμα. Είναι η επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που έμειναν μέχρι αυτή την ώρα, ακόμα και αν είναι λίγοι, της Επιτροπής Πολιτισμού και τους ε, ε, πάρα πολλούς βοηθούς και συνεργάτες που δεν μας άφησαν στη μοναξιά μας. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.